Ja, guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Είναι η ώρα 9 και 10. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Στο σημείο 1 της ημερησίας διάταξης έχω δύο ε, ανακοινώσεις, μία μάλλον. Το σημείο 18, η έκθεση Γκαρντίνη δεν προβλέπεται, προβλέπεται κανονικά για Πέμπτη η ε, στις 10, αλλά θα αναβληθεί για τις 19 Σεπτεμβρίου. Θα... θα σας ενημερώσουμε όλους σχετικά με το τι ώρα θα ξεκινήσουμε την εξέταση της ημερήσιας διάταξης ε, την Πέμπτη. Θα σας ε, στείλουμε πολύ σύντομα email. Σημείο 2 της ημερησίας διάταξης. Ε, έχουμε διερμηνία. Έχουμε διερμηνία και στα εσθονικά, λετωνικά και κροατικά, κροατικά μόνο για την Πέμπτη. Έχουμε επίσης σε μια ομάδα επισκεπτών από την Ιταλία που βρίσκονται, δεν έχουν έρθει ακόμα φαίνεται. Θα τους καλωσορίσουμε αργότερα λοιπόν. Και Έχουμε μοιράσει μια έκθεση στους ε, συναδέλφους σχετικά με την επίσκεψη της ΕΦΣΑ. Ε, στα έγγραφά σας υπάρχει αυτή. Και να καλωσορίσω και ένα νέο μέλος της Επιτροπής μας, παλαιός γνωστός. Πρόκειται για τον συνάδελφο Τόμα Σούλμερ ε, από το ΕΛΚ που θα ξαναεργαστεί μαζί μας ως πλήρες μέλος τον ε, συγχαίρουμε, δεν τον βλέπω ακόμα όμως ε, και έχουμε ένα νέο αναπληρωτή, τον συνάδελφο Έρικ Μπανκή από την Ουγγαρία. Είναι Ευρωβουλευτής από την 1η Ιουνίου. Σας καλωσορίζουμε θερμά στην Επιτροπή μας. Ε, στην καλή συνεργασία μαζί σας. Άλλη μία Ανακοίνωση, έχουμε μια έκθεση για την ε, ανακύκλωση. Όλα τα στοιχεία, τα σχετικά θα τα βρείτε στα έγγραφά σας. Ε, και παρακαλώ να φέρετε τα έγγραφα σας και την επόμενη φορά για να μην χρειάζεται να τα ξαναμοιράσουμε για να κάνουμε οικονομία στους πόρους. Φτάνουμε έτσι στο σημείο 3 της ημερησίας διάταξης Πρόκειται ε, για την ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων. Ε, Η συγητής, ο συνάδελφος Μύροσλαβ Ούσκι. Μύροσλαβ, ε, παρακαλώ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, θα ήθελα να σας μιλήσω όσο πιο καθαρά γίνεται και γι' αυτό διάλεξα να μιλήσω τσέχικα. Περιμένω για να έχουν όλη την ευκαιρία να φορέσουν τα ακουστικά τους, ούτως ώστε να με καταλαβαίνουν όλοι καλύτερα. Σκοπός της έκθεσης και των ε, τροπολογιών είναι να προσαρμοστεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις τεχνικές εξελίξεις όσον αφορά τις τεχνικές ε, δοκιμές. Και αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε το θόρυβο ολιστικά, σφαιρικά, σαν ένα γενικό πρόβλημα. Υπάρχουν διάφορες πηγές θορύβου, επιφάνεια των δρόμων, ελαστικά, ε, κινητήρες. Είναι συνδυασμός διαφόρων ε, παραγόντων. Τώρα στις τροπολογίες υπάρχουν διαφορές μεταξύ μονίμων ε, επιτροπών, μεταξύ πολιτικών ομάδων όσον αφορά την ετικετοθεσία. Όπως έχουμε δεσμευτικούς κανόνες για τα επίπεδα εκπομπών σε γραμμάρια ε, διοξιδίου του άνθρακος, λοιπόν όπως έχουμε ετικετοθεσία και για τις εκπομπές ρήπων, τώρα έχουμε και το θέμα κάποιες ετικετοθεσίες όσον αφορά το θόρυβο. Νομίζω ότι ο θόρυβος, το επίπεδο θορύβου πρέπει να υπόκειται σε αξιολόγηση ε, αντιχτύπου και αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω υποβάλει την τροπολογία 33 που θέλει να θεσπιστεί ένα σύστημα ταξινόμησης οδικών των επιφανειών των δρόμων, ούτω ώστε να μπορούμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ επιφανειών που είναι πιο ήσυχε και άλλων που παράγουν περισσότερο θόρυβο. Από την ε, άποψη της ε, ανθρώπινης υγείας, ε, μου δημιουργείται ένα πρόβλημα όσον αφορά τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά οχήματα. Να εξετάζονται ξεχωριστά. Νομίζω ότι οι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα οχήματα. Κάποιες τροπολογίες αναφέρονται στην ταξινόμηση διτρόχων και τριτρόχων οχημάτων, μοτοσυκλετών και τριτρόχων αυτά είναι θέματα που δεν εμπίπτουν σε αυτή την νομοθεσία ε, και εγώ είμαι υπέρ ξεχωριστής αντιμετώπισης των μοτοσυκρετών σε ξεχωριστή νομοθεσία. Η κατηγορία νη 1 είναι φορτηγάκια και οχήματα υπάρχουν μόνο σε μερικά κράτη-μέλη και υπάρχουν και σχετικές τροπολογίες για αυτά τα οχήματα. Μιλάμε για οχήματα που έχουν κινητήρα κάτω από 600 κυβικά εκατοστά. Πολύ συχνά είναι τα μικρά οχήματα που, για το, που μοιράζουν οι γαλατάδες στο γάλα και υπόκειται στους κανόνες ένα και δεν θα έπρεπε να εμπίπτουν στην συγκεκριμένη νομοθεσία διότι δεν υπάρχει άλλη πηγή θορύβου από αυτά τα οχήματα. Ε, υποστηρίζω και τις τροπολογίες που αφού αφορούν τους μικρούς κατασκευαστές, τους κατασκευαστές μικρής κλίμακας, με μικρή παραγωγή, μικρό, χαμηλό αριθμό οχημάτων. Πιστεύω θα πρέπει να εξαιρούνται από αυτή την ομοθέσια. Ξέρω ότι η ομάδα S&D ε, ζητά πληροφορίες, ζητά ενημερωτικό υλικό για το θορύβους. Ε, τα, τα ενημερωτικά έντυπα για τα θέματα θορύβου είναι διαθέσιμα στα σημεία πώληση οχημάτων. Θα ήθελα οι κατεξουσιοδότητες συμπράξεις να περιοριστούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί διάφορα επιχειρήματα που σχετίζονται με την οξύ ανάγκη για τεχνικές αλλαγές. Δεν κατανοώ πραγματικά πώς ο θόρυβος των κινητήρων θα μας οδηγεί σε μια κατάσταση όπου ξαφνικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εξαιρεθεί από τις διαδικασίες λήψης απόφασης. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Έχουμε και το παράτημα 3, το οποίο καλύπτεται από την έκθεσή μας. Αφορά τις οριακές τιμές. Είμαι υπέρ μακροπρόθεσμης τέταρτης φάσεως. Ξέρω ότι δεν συμφωνούν όλοι με την τέταρτη φάση. Όμως α, θα σας έλεγα ότι και στην άλλη νομοθετική δουλειά που κάνουμε σκεφτόμαστε πολύ μακριά στο μέλλον. Καμιά φορά βλέπουμε τι θα γίνει και σε μία εικοσαετία και δεν καταλαβαίνω γιατί ο θόρυβος των οχημάτων θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες που αφορούν το παράρτημα. Θα έπρεπε να σας πω παρεμπιπτόντως ότι έχουμε 146 τροπολογίες συνολικά. Και το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αν θέλουμε να έχουμε συμβιβασμούς βάσει συνενέσους θα πρέπει να αφιερώσουμε πολύ προσοχή στο παράρτημα 3. Αυτό θα είναι και το δυσκολότερο σημείο. Γι' αυτό το λόγο και για άλλους λόγους εγώ θα σας πρότεινα να αναβάλουμε την ψηφοφορία για το σημείο αυτό από την τελευταία συνεδρίαση πριν τις διακοπές και να το συζητήσουμε στην πρώτη συνεδρίαση μετά τις θερινές διακοπές. Κι άλλο ένα επιχείρημα που υποστηρίζει κάτι τέτοιο είναι ότι το Συμβούλιο δεν ξεκίνησε ακόμα επεξεργασία του ζητήματος και τακτικός πώς δεν είμαι πεπισμένος ότι θα έπρεπε απαραίτητα να έχουμε θέση του Κοινοβουλίου αμετακίνητη πολύ νωρί όταν δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι η θέση του Συμβουλίου. Αυτό αποτελεί μόνο μια δική μου σύσταση. Ε, δεν είναι κάτι το οποίο θα σας πιέσω να το δεχτείτε, αλλά θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η άποψη των σκιωδών εισηγητών επ' αυτού. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω να τα καταφέρουμε να μειώσουμε την ηχορύπανση από τα οχήματα, ούτως ώστε να βελτιώσουμε και την ανθρώπινη υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ κύριε Μυροσλάβ Ούσκι. Ε, είναι μια κατάσταση που βλέπουμε συχνά, ασκούμε ασκούν πίεση στο Κοινοβούλιο να κάνουμε τη δουλειά μας γρήγορα, αλλά τη δουλειά μας εμείς την έχουμε τελειώσει. Ε, το Συμβούλιο αργεί. Εμείς ε, τρέχουμε σαν τεζεβέ, ενώ το Συμβούλιο τρέχει σαν καρβουνιάρης. Και αυτό πολύ συχνά μπλοκάρει τις εργασίες ε, στην νομοθετική διαδικασία. Αλλά αυτό ίσως ε, θα έπρεπε να το συζητήσουμε στον κατάλληλο, στον κατάλληλο χώρο. Ε, Σκιώδης ηγητής είναι ο κύριος Ταρταρέλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάνω απ' όλα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ούσκι για την καλή δουλειά που έκανε και επειδή ε, δέχτηκε πολλές από τις δικές μου τροπολογίες πιστεύω ότι έκανε ένα έγγραφο, ετοίμασε ένα πολύ συνεκτικό έγγραφο παρά το θέμα που δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο είναι αρκετά τεχνικό και πολύ πολιτικό στη φύση του. Στη δέσμη τροπολογιών μου προσπάθησα να διευκρινίσω τη θέση μας. Θα σταθώ μόνο σε κάποια σημεία. Ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόβλημα μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, σφαιρική. Δεν θα ήθελα δηλαδή όλη προσπάθεια για τη μείωση των θορύβων να επικεντρώνεται μόνο στους κινητήρες και στα αυτοκίνητα. Ο θόρυβος είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Είναι και αποτέλεσμα παραδείγματος χάρη και της συμπεριφοράς του ανθρώπου, αλλά και πάνω απ' όλα των οδικών υποδομών. Επ' αυτού υπάρχει λίγη προσοχή που έχει δοθεί στο θέμα αυτό από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ζητάμε σε μια προσέγγιση οριζόντια και ολοκληρωμένη να ακολουθηθεί για το πρόβλημα. Να αναλάβει την όλη προβληματική λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προβλέψει επί τη ευκαιρία των νέων προγραμμάτων για τα διαθωτικά ταμεία να προβλέψει κάποιες, κάποιους προσανατολισμούς ώστε να επιτραπεί στα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την κατάσταση των οδοδρόμων κυρίως εκείνων των δρόμων με μεγάλη κυκλοφορία των μεγάλων πόλεων πάνω απ' όλα. Στις τροπολογίες υπάρχουν και κάποιες ε, ενδείξεις που εξέφρασε τέλεια ο κύριος Ούσκι σε θέματα ταξινόμησης των οχημάτων όπως και ε, ο πινακίδα για τη μείωση των, ε, ο πίνακας για τη μείωση των δεσιμπέλ. Θα πρέπει να προσέξουμε κάποια οχήματα που είναι πολύ γρήγορα και με παράγονται σε μικρούς αριθμούς. Στους πίνακες λοιπόν που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά τα οχήματα έχουν τοποθετηθεί μαζί με άλλα οχήματα που παράγονται σε μεγαλύτερο αριθμό και κυκλοφορούν περισσότερα από αυτά. Όμως αυτά εκπροσωπούν μόνο μία παραγωγή 0,03% της συνολικής αγοράς της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη. Για αυτή την ιδιαιτερότητά τους εγώ θεώρησα ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια άλλη ε, κατηγορία και θα παρακαλούσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσέξει δεόντως το θέμα αυτό και να δεχτεί αυτή την πρόταση γιατί μιλάμε για οχήματα που είναι εντελώς διαφορετικά από όλα τα άλλα και στην τροπολο... στις τροπολογίες ε, αναφέρω και κάποια πολύ τεχνικά ζητήματα και συμφωνώ με τον εισηγητή. Ε, δύο μέτρα ένα δευτερόλεπτο και όχι τρία μέτρα ένα δευτερόλεπτο να χρησιμοποιήσουμε που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις δοκιμές. Και κάτι που είναι πολύ σημαντικό και το προτείνει και η συνάδελφος η Άνια το θέμα της ετικοτασίας, του labeling. Εγώ είμαι υπέρ ε, αυτής της διαδικασίας η ΠΕΡ είναι χρήσιμη κυρίως για τον καταναλωτή που τη στιγμή της επιλογής θα πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία στη διάθεσή του για να μπορεί να κάνει μια επιλογή ε, ενήμερος ε, και να κάνει μια αποδεκτή και βιώσιμη επιλογή. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μεθοδολογικό πρόβλημα. Δηλαδή, α, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια επιλογή και χρειάζεται μια διαδικασία συνέπειας και ε, συνεπιών και μια ad hoc διαδικασία για το labeling. Και να μην περιορίσει την Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στο πρόβλημα αυτό, αλλά η θέση μου είναι ότι θα πρέπει να μετατεθεί σε μεταγενέστερο στάδιο χρονικά και εγώ θα έλεγα ότι το θέμα του labeling σε αυτή τη φάση θα μπορούσε να είναι κάτι επιζήμιο κυρίως για, τις μικρές, για τα μικρά οχήματα. Δηλαδή, εκείνα που κοστίζουν λιγότερο στην αγορά. Κάτω των 10.000 ευρώ σε κόστος. Σημαντικό κομμάτι της αγοράς και για ε, χρήση που δεν είναι πολύ σημαντική οικονομικά. Λοιπόν, να φορτωθούν το βάρος της διαδικασίας αυτής νομίζω ότι είναι κάτι εντελώς άδικο, άρα θα ήθελα να το προσέξουμε αυτό. Ε, μήπως εισάγει αυτή η νομοθεσία έτσι βία στην οδηγία χωρίς να γίνει εξολόγηση συνεπιών θα μπορούσε να δημιουργήσει στρεβλώσεις όσον αφορά την πρόσβαση στις μεγάλες πόλεις, στα ιστορικά κέντρα κλπ. των οχημάτων. Είναι σειρά σημαντικών ζητημάτων, πολύ ευαισθητών, που θα πρέπει να συζητηθούν ε, δεόντως. Τελευταία πτυχή που θα ήθελα να αναφέρω στον αφορά το δεξίδιο του Άνθρακος. Είναι ένα θέμα με το οποίο συχνά ασχολούμεθα σε αυτή την ε, επιτροπή. Η τεχνολογία έκανε γιγαντία βήματα. Κάθε μέρα κάνει βήματα στην προσπάθεια μείωση εκπομπών, θορύβων κλπ. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις πρόοδους. Όμως θα πρέπει να προσέξουμε ένα στοιχείο. Κάθε συμπίεση μεγέθους του, του κινητήρα ε, δημιουργεί αύξηση βάρους τελικά ε, γενικά το οχήματο και οδηγεί σε μεγαλύτερη εκπομπή ε, ε, του, εξοδείου εξοδίου του άνθρακος. Εκτιμώ τη δουλειά που έκανε ο εισηγητής, το λέω ξανά, και όσον αφορά την ψηφοφορία στην Επιτροπή, και εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να, το, να κάνουμε ψηφοφορία το Σεπτέμβριο αντί τον Ιούλιο. Αυτά και ευχαριστώ. Eh, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ κύριε Σιγητά, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι καλή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία τροποποιεί τον υπάρχοντα μηχανισμό. Συμφωνώ όμως με τους συναδέλφους που λένε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες. Δεν υπάρχει μόνο ο θόρυβος ε, του κινητήρα. Υπάρχουν ε, και άλλοι παράγοντες που δημιουργούν η χορύπανση. Πολλές φορές ο θόρυβος είναι κάτι που δεν ε, ακούγεται και πολύ αν μπορώ να πω. Και είναι περίεργο αυτό. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να εντάσσονται στο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Θα πρέπει να δούμε τα ελαστικά και πολλούς άλλους παράγοντες. Στην οδηγία αυτή βλέπουμε ότι ε, η εστίαση γίνεται στα οχήματα και στο θόρυβο. Αλλά δεν γίνεται ουσιαστικά, δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το ζήτημα της διαχείριση της κυκλοφορίας. Αλλά πρέπει αυτό το ζήτημα να λυθεί και να το πραγματεύεται και η επόμενη οδηγία που θα εκπονηθεί. Δεν έχουν γίνει όμως τα δέοντα κατά την άποψή μου. Είναι λίγα αυτά που προβλέπονται μέχρι στιγμής. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και η ελάχιστη, ε, κατώτα τουλάχιστη υποχρεωτική ελαστικότητα και ευελιξία. Υπάρχει η πρόβλεψη για τη μείωση των δεσιμπέλ μέσα σε 10 χρόνια, μήπως θα έπρεπε όμως να υπάρχουν κάποια στάδια για τους ε, κατασκευαστές. Να υπάρχει μια μεταβατική περίοδο. Σίγουρα οι στόχοι της οδηγίας όμως θα πρέπει να είναι φιλόδοξοι, άρα πρέπει να τροποποιηθεί το σχέδιο. Επαναλαμβάνω ότι καλό θα ήταν να υπάρχουν κάποιοι ενδιάμεσοι στόχοι κάποια διάμεσα στάδια. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να προβλέψουμε παρεκκλήσεις για τα αθλητικά, για τα σπορ οχήματα. Υπάρχουν άλλες κατηγορίες οχημάτων που ρηπαίνουν, που ήχο ρηπαίνουν πολύ περισσότερο και δεν λαμβάνονται υπόψη. Και οι μέθοδοι τεστ δοκιμών και τα labels. Ο συνάδελφος το ανέφερε, το έχουμε συζητήσει. Πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα επισήμανσης Έχουμε την περιβαλλοντική απόδοση, το, την ηχοστάθμη, όλα αυτά που να λαμβάνονται υπόψη. Και καλό θα ήταν να γίνει και μία μελέτη. Βέβαια αυτό παίρνει χρόνο. Όχι όμως, να μην γίνει αυτό τρία χρόνια μετά, γιατί αυτό προβλέπεται στο παράρτημα 3 πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύω τη οδηγία. Αυτό θα πρέπει να λέγεται. Και όχι τρία. θα ολοκληρώσω με την εξή σκέψη. Η οδηγία, το σχέδιο οδηγίας είναι καλό, αλλά μπορεί να βελτιωθεί. Επίσης μπορούν να δοθούν μεγαλύτερα περιθώρια στον κλάδο της βιομηχανίας για να πετύχουν τους στόχους. Ουσιαστικά δηλαδή πρέπει να ορίζουμε το στόχο και όχι τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί αυτός. Και παραλαμβάνω τον αριθμό των παρεκκλήσεων θα πρέπει να το περιορίσουμε. Ο κοινό είναι ο στόχο να μειωθεί η μα Και αν μου επιτρέπετε να πω κάτι τελευταίο για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι θέλουμε να προσθέσουμε ουσιαστικά θόρυβο. Και αυτό βέβαια αντιβαίνει και το στόχο. Όταν κάποιο αγοράζει ένα ηλεκτροκίνητο όχημα, έχει κάποιο στόχο που εδώ δεν ε, λαμβάνουμε Σας ευχαριστώ πολύ, ε, ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα ε, επιχειρήματα σχετικά με την έκθεση του κυρίου Ούς εγώ δεν πιστεύω ότι η Κομισιόν έχει υποβάλει καλή πρόταση διότι προτείνει η κατηγοριοποίηση οχημάτων ε, που καθόλου δεν ανταποκρίνονται ε, στα πρότυπα της εποχής μας. Αυτό μεταξύ το έχει ε, παραδεχτεί η Κομισιόν. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ καλή η διαδικασία της συναπόφασης για να ρυθμίζονται τα πράγματα που δεν έχει κάνει πολύ καλά η Κομισιόν. Ο εισηγητής ε, προτείνει τρόπο κατηγοριοποίησης που κατά τη γνώμη μου μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητάμε. Ε, αντιστοιχεί στο, στην σχετική κατηγοριοποίηση των ε, οχημάτων και πιστεύω ότι αυτή την κατηγοριοποίηση θα πρέπει να πάρουμε ως βάση. Ο πυρήνας αυτού του κανονισμού βρίσκεται στο παράρτημα 3. Έχουμε ένα σωρό τροπολογίες. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Ε, θα πρέπει να εξετάσουμε το εξή πιο προσεκτικά αν θέλουμε να καταλήξουμε σε συμβασμό. Τροπολογίες ε, που προτείνουν ε, όρια για γιοταχή, είτε μιλάμε για οχήματα σπόρη, είτε για κανονικά του δρόμου και που προτείνουν όρια κάτω των 60 δεσιμπέλ. Αυτό δεν είναι εφικτό, οπότε δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοια όρια. Τα ηλεκτρικά οχήματα δεν κάνουν ε, θόρυβο. Ε, που, δεν κάνουν θόρυβο που ακούγεται. Ε, αυτά έχουν ηχοστάθμη 67 δεσιμπέλ. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν τα βενζινοκίνητα οχήματα να τα φέρουμε πιο κάτω από το όριο αυτό. Δεν υπάρχει τεχνικός τρόπος να επιτευχθεί αυτό. Γι' αυτό για μένα είναι σαφές ότι εγώ δεν πρόκειται να βάλω την υπογραφή μου σε κανένα παράρτημα 3 όπου να υπάρχουν οριακές τιμές μέχρι 67 δεσιμπέλ. Ούτε καν με προθεσμία 5 ετών. Ε, αυτό δεν είναι εφικτό. Έτσι θα ε, νομοθετήσουμε, ε, θα φτιάξουμε ένα νόμο ο οποίος δεν είναι σκόπιμος. Η όλη συζήτηση δεν είναι σκόπιμη ας ε, θέσουμε οριακά, οριακές τιμές οι οποίες ε, να είναι ρεαλιστικές. Επίσης ε, θα πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και όσον αφορά την επισήμανση θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι εάν υπαγορεύσουμε ένα τέτοιο σύστημα επισήμανσης στην νομοθεσία, τότε θα πρέπει ε, να είναι μια επισήμανση που να ενημερώνει τον ε, αγοραστή, τον καταναλωτή. Ε, κάτι που δεν λειτουργεί όμως είναι Ε, η σφραγίδα πάνω στο αυτοκίνητο που λέει ότι το αυτοκίνητο αυτό ε, δεν κάνει πολύ ε, θόρυβο. Αυτό έχει να κάνει με την άδεια κυκλοφορία του αυτοκίνητου. Αυτό μπορεί να είναι εντάξει, αλλά δεν έχει θέση στη συγκεκριμένη πρόταση. Πρότεινα να διαγραφούν οι ελάχιστες απαιτήσεις, θα σας πω γιατί σύντομα δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες σχετικά με το πότε είναι υπερβολικά ήσυχα ε, τα οχήματα. Και πιστεύω ότι αυτό το θέμα δεν έχει θέση σε έναν κανονισμό που έχει να κάνει με το περιβάλλον. Αυτό είναι θέμα ασφαλείας ε, των οδικών ε, μεταφορών. Και τρίτον, προτάσεις προαιρετικού χαρακτήρα, θελοντικού χαρακτήρα ε, δεν έχουν κανένα νόημα. Εάν ε, θέλουμε να νομοθετήσουμε τότε ε, εμπεριστατωμένα και όχι με τον τρόπο αυτόν. Και μία προτελευταία παρατήρηση Ακούω πάντα ευχαριστώ στον κλάδο των αυτοκινήτων, τη βιομηχανία των αυτοκινήτων ε, και είμαι διατεθειμένος ε, στην διαδικασία να ε, υποβάλω τροπολογίες εάν οι τροπολογίες αυτές είναι περιστατωμένες. Δεν είμαι διατεθειμένος όμως να συμμετάσχω σε αυτό το πάρτι των τροπολογιών, τον χαρτοπόλεμο, χωρίς να γίνει μια καλή συζήτηση. Γι' αυτό δεν έχουμε συνυπογράψει όλε αυτέ τι τροπολογίε. Ευχαρίστω θα κάτσω να ακούσω ε, τι προτεραιότητε που υπάρχουν ε, και ε, σωστή επιχειρηματολογία. Αλλά αυτόν τον χαρτοπόλεμο των τροπολογιών, όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο, δεν μ' αρέσει, δεν έχω συμμετάσχει σε αυτό και γι' αυτό δεν έχω συνυπογράψει τις τροπολογίες αυτές, γιατί δεν πιστεύω ότι όλες έχουν, τροπολο... έχουν προτεραιότητα, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο παράτημα 3. Τελευταία παρατήρηση, το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Όσον αφορά την τεχνική νομοθεσία, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τον χρόνο ώστε να κάνουμε ποιοτική δουλειά και ε, μήπως θα ήταν γι' αυτό σκόπιμο να ψηφίσουμε μετά το καλοκαίρι από το Συμβούλιο άκουσα όμως ότι αυτοί μας πετάνε εμάς τον παλάκι και λένε θα ξεκινήσουν αφού ολοκληρώσει το Κοινοβούλιο. Ε, θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ε, να μην ε, γίνεται αυτή η δουλειά με το Συμβούλιο να κατηγορεί ο ένας τον άλλον και να θεωρεί ότι είναι ευθύνη του άλλου η καθυστέρηση, αλλά θα είναι σημαντικό να έχουμε τελικά ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ισά του Χάση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά του. Δουλειά που έκανε για την Επιτροπή μας. Διάφορα στοιχεία που προτείνει ο εισηγητής ε, είναι σημεία επί των οποίων συμφωνώ και τα υποστηρίζω, όπως η ενημέρωση των καταναλωτών. Όμως ε, δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιες, κάποιες παρατάσεις που ζητά ο εισηγητής στον αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Πέρασε πολύ καιρό μετά τον καθορισμό των οριακών τιμών για τα οχήματα και όλοι γνωρίζουμε ε, πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι ο περιβαλλοντικός θόρυβος και τι δυσκολίες δημιουργεί για πολλούς ανθρώπους. Μία μείωση θορύβου κατά ένα δεσιμπέλ κοστίζει περίπου 0,5% του κόστους ενός αυτοκινήτου. Τα ωφέλη όσον αφορά την υγεία που επιτυγχάνονται με αυτή τη μείωση, δηλαδή όταν ο κόσμος κοιμάται καλύτερα και ασθενεί λιγότερο, είναι αρκετά ξεκάθαρα. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι οικονομικά είναι 30 φορές πιο επωφελές, έχεις 30%, 30 φορές περισσότερη, περισσότερο ωφέλη όσον αφορά την υγεία από αυτή τη μείωση. Άρα δεν πρέπει να θεωρείται ένα οικονομικό άχθος. Γι' αυτό δεν είμαι υπέρ της παρατάσεως προθεσμιών. Ήδη υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα που πληρούν τις οριακές τιμές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις δικές μου τροπολογίες προσπαθώ να καθορίσω οριακές τιμές για δίτροχα και τρίτροχα αυτοκίνητα, οχήματα. Είμαι επίσης υπέρ μειώσεως ε, των οριακών τιμών και είμαι υπέρ ξεχωριστής, ξεχωριστών ορίων μάλλον όσον αφορά το χρονικό ορίζοντα 2020 όπως είπαν οι συνάδελφοι, δεν μιλάμε μόνο για το θόρυβο των κινητήρων, μιλάμε για την επιφάνεια των δρόμων και για το θόρυβο που παράγουν τα ελαστικά. Αυτό που θα πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας είναι ότι θα, δεν θα έπρεπε να ρίχνουμε τον μπαλάκι σε άλλους. Δεν θα ήταν ενδεδειγμένο εμείς να εθελοτυφλήσουμε όσον αφορά τους θορύβους των κινητήρων με το επιχείρημα ότι τα ελαστικά επίσης παράγουν θόρυβο. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αποφεύγουμε χειραγώγηση και διάφορα κόλπα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι όταν μετρούμε τον θόρυβο παράγουν τα οχήματα θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί τα πιο θορυβόδια ελαστικά στα χήματα αυτά. Οπότε θα είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί ο θόρυβος των λαστικών για να αλλάξει αποτελέσματα. Ευχαριστώ κυρία Βίλς. Ευχαριστώ πολύ. Ο θόρυβος ε, από την ε, κυκλοφορία ε, είναι πανταχού παρόν στις πόλεις μας και μαζί με τις εκπομπές αερίων των ε, αυτοκινήτων ε, είναι και ο θόρυβος ε, κάτι που επιβαρύνει την υγεία των ανθρώπων. Και σημαντικό είναι ότι το στρες προκαλείται όχι μόνο από δυνατό θόρυβο για σύντομο χρονικό διάστημα, ο εγκέφαλος ε, συνεχώς επεξεργάζεται τους ε, ήχους του περιβάλλοντος ακόμα και κατά τον ύπνο. Ε, περισσότερα δεσιπέλ, κυρίως κατά τις περιόδους ανάπαυσης, σημαίνει περισσότερο στρες για τους ανθρώπους, επιβάρυνση του σώματος και αύξηση της, της πίεσης. Μείωση λοιπόν του θορύβου θα σημάνει σημαντική βελτίωση ε, του βιωτικού επίπεδου των ανθρώπων. Ε, γι' αυτό αξίζει τον κόπο να κάνουμε κάτι εδώ και να μειώσουμε τον ε, θόρυβο από την κυκλοφορία. η πρόταση του εισηγητή ε, να αποδυναμώσει τόσο πολύ τα, ε, τις οριακές τιμές ε, και να αναβάλει την, την εφαρμογή του σε επάπειρον, αυτό δεν νομίζω ότι είναι πολύ καλό. αναφέρεται σε μείωση κατά ένα δεσιμπέλα αλλά είναι απίστευτη η προσέγγιση αυτή. Εμένα μου θυμίζει τον κανονισμό για την ε, μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα των αυτοκινήτων. Τότε ε, ο βιομηχανικός τομέας ήθελε να, ε, αυξηθούν οι ανώτατες τιμές, να είναι πιο ήπιες οι τιμές δηλαδή, και Μάλιστα, η, ε, η, διάφοροι ε, κατασκευαστές ε, έχουν υποβάλει τις δικές τους προτάσεις, αλλά εγώ θα ήθελα να καλέσω τους συναδέρφους να μην ακολουθήσουν τις εκκλήσεις των κατασκευαστών. Δεν είναι απαραίτητο όμως ε, να προσαρμόσουμε τις ανώτατες τιμές, διότι ε, ήδη οι περισσότεροι κατασκευαστές ήδη πληρούν ε, τις προϋποθέσεις της φάσης 1. 70 δεσιμπέλ δηλαδή μέχρι το 2014 ε, και πολλοί επίσης ε, πληρώνουν ε, τη φάση 2, 68 δεσιμπέλ μέχρι το 2020. Υπάρχουν λύσεις, απλά θα πρέπει να εφαρμοστούν. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με το συμφέρον των ανθρώπων. Γι' αυτό θέλουμε πιο σύντομη ε, εφαρμογή ε, της πρότασης της Κομισιόν. Θέλουμε την ε, πρώτη φάση μέχρι το 2013 και την δεύτερη φάση μέχρι το 2015 και θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ένα τρίτο βήμα μέχρι το 2020 όπου θα εξετάσουμε περισσότερο τα φορτηγά. Παρότι μόνο το 3% όλων των οχημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι φορτηγά, αυτά προκαλούν το ε, ε, μισό των ε, εκπομπών. Και η Κομισιόν έχει δίκιο που λέει ότι και το επίστρωμα του δρόμου παίζει ρόλο κατά το θόρυβο, αλλά πιο είναι όμως ταυτόχρονα και ο πιο απλός τρόπος να μειώσουμε τον θόρυβο. Ε, εδώ όμως μιλάμε για ε, κανονισμό για τις μηχανές των αυτοκινήτων ε, και όχι για τα επιστρώματα των οδών. Ο κύριος Ρώση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή όσον αφορά τη σήμανση, το label, τη δυνατότητα παρατάσεων αλλά τέτοιες στιγμές νομίζω ότι είναι αδύνατο να ζητήσουμε πολλά από τους κατασκευαστές. Η αγορά καταραίει συνεχώς, φτάνει να δούμε τους οικονομικούς δείκτες και στι τελευταίε μελέτες και εξακολουθούν να ζητούμε, το να ζητούμε θυσίες σε αυτές τις στιγμές κινδυνεύουμε με μετεγκαταστάσει, κλεισίματα κλπ. και απώλεια θέσεων εργασία. Θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα όσον αφορά τα αποτέλεσμα που επιτυγχάνονται όταν ζητάμε πολλά. Στην Ιταλία ε, είχαν τεθεί πολύ χαμηλά όρια στους Σήμερα Κανένα, κανένας κατασκευαστές δεν μπορεί να σεβαστεί αυτά τα όρια. Δεν υπάρχουν κινητήρες παρά τις προσπάθειες μειώσεως του ρίβου που να μην ξεπερνάνε τα όρια αυτά. Οπότε όλες οι κοινότητες Ιταλίας κάθε φορά ε, ε, δίνουν παρέκκληση κάθε φορά. Αυτά ήταν όρια που είχα τεθεί για τις ε, οικοδομές. Και κάθε φορά πρέπει να δίνουν παρεκκλήσεις οι κοινότητες γιατί είναι αδύνατο να μην ξεπεραστούν τα όρια θορύβου για τις ε, οικοδομές. Άρα γίνονται κάθε φορά ασκήσεις ε, άχρηστες, ύφους, πολιτικές. Λοιπόν, και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που προτείνει ο εισηγητής τελικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχω πρόβλημα. Εφτά έχουν ζητήσει το λόγο. Ε, Έχουμε λοιπόν 7 ομιλητές στον κατάλογο και έχουμε μετά και την έκθεση του Ζιλ Παρνιό. Γι' αυτό θα πρέπει να περιορίσω σε 1,5 λεπτό τον χρόνο ομιλίας ώστε να προλάβουν όλοι να πάρουν το λόγο. Η συνάδελφος Βάις Γκέρμπερ, ε, που είναι η συγγήτρια στην ε, Επιτροπή ε, Ενιαίας Αγοράς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον ε, εισηγητή κύριο Ούσκι. Η ΙΜΚΟ θα ψηφίσει αυτή την εβδομάδα, έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά Έχουμε ασχοληθεί πολύ και με το παράρτημα 3 και ε, τις προτάσεις που είναι σημαντικές ε, για τους καταναλωτές. Έχουμε ε, ολοκληρώσει τις εργασίες μας, έχουμε καταλήξει σε συμβιβασμό μεταξύ των πολιτικών ομάδων και με εκπλήσει η αναβολή, διότι εμείς καταβάλαμε κάθε προσπάθεια ώστε να τηρήσουμε αυτό το πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα και τα καταφέραμε. Και τώρα παρόλα αυτά έχουμε αναβολή. Αλλά τέλος πάντων... Ε, δεν θα σας κάνω τη ζωή δύσκολη. Όσον αφορά τα όρια της, του θορύβου, είναι σημαντικό για λόγους υγείας να μειωθεί το επίπεδο θορύβου. Στηρίζω το ότι έχουμε μακροπρόθεσμους στόχους. Στην έκθεσή μου στην ΙΜΚΟ έχω προτείνει ε, μακροπρόθεσμου μακροπρόθεσμους στόχους. Ε, η ε, Κομισιόν προτείνει δύο βήματα μετά από δύο και μετά από πέντε χρόνια. Ε, πιστεύω ότι είναι σημαντικό και για τους καταναλωτές να έχουμε και μακροπρόθεσμο στόχο, ο οποίο να είναι φιλόδοξο. στον ε, συνάδελφο Κράμερ να πω ότι δεν βρίσκω καλή την πρόταση ε, της Κομισιόν ε, για τις κατηγορίες. Δεν είναι αρκετά διαφοροποιημένη και επίσης πεπαλαιωμένη είναι η πρόταση αυτή. Σε κάποιες από τις κατηγορίες αυτές δεν υπάρχουν πια αυτοκίνητα. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε άλλη κατηγοριοποίηση. Έχω εκπονήσει εγώ μια σχετική στην ΙΜΚΟ, διότι είναι δυνατή η διαφοροποίηση αλλά χρειάζεται να είναι πιο ρεαλιστική και πιο φιλόδοξη από την πρόταση της Κομισιόν. Ε, χρειαζόμαστε όμως και πιο ρεαλιστικούς στόχους από αυτούς της Κομισιόν. Ε, η συνάδελφο Βίλη είπε ότι έχουμε την ίδια συζήτηση με το διοξίδιο του άνθρακα. Ε, ο βιομηχανικό τομέα συζητά από εμά να κάνουμε πιο ήπιε τι διατάξει. σύντομα, σε σύντομη θα είμαι. δεν θέλουμε να διακυβεύσουμε και τους στόχους σχετικά με, την, ε, με τις εκπομπές ε, του διοξιδίου του άνθρακα. Βρίσκω σημαντική και την ενημέρωση των καταναλωτών. Δεν χρειάζεται όμω ε, να το συμπεριλάβουμε αυτό στο σχετικό κανονισμό. Ευχαριστώ πολύ, ο Ρίχαρτ Σέμπερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι σημαντικό, σημαντικό επιχείρημα εδώ είναι η προστασία της υγείας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να πούμε ότι η ολιστική αυτή προσέγγιση που ζητούν οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι σωστή. Και γι' αυτό τίθεται και το θέμα αν πρέπει να είμαστε τόσο φιλόδοξοι όσο ε, είναι οι συνάδελφοι. Σημαντικό είναι να ασχοληθούμε με το θέμα του θορύβου και τις επιπτώσεις στην υγεία. Αλλά ε, είπαμε ότι τα επιστρώματα των οδών είναι ε, πολύ σημαντικός παράγοντας, ιδιαίτερα στις υψηλές ταχύτητες. Υπάρχουν και μεγάλες διαφορές ανάμεσα στην ποιότητα των επιστρωμάτων και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις θέσεις ε, των συναδέρφων, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για το παράρτημα 3 διότι ε, εδώ έχουμε συνθήκες οι οποίες δεν ε, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Επίσης ε, θα πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να... Ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην ε, έχουμε αρνητικές συνέπειες ως προς το κόστος των αυτοκινήτων με τις διατάξεις αυτές. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε γενικά το θέμα του θορύβου, διότι υπάρχουν πολλές μικρές πηγές θορύβου οι οποίες συσσωρεύονται και που οδηγούν σε προβλήματα για τους ανθρώπους. Ε, χρήσιμο είναι να έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση. Γενικά όμως νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ε, ε, κατά νου τη συνολική εικόνα. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Ρίχαρτ Τζίπερ, ο Καλχάτς Φλόρενς. ευχαριστώ. Ναι, πάλι είμαστε στο αγαπημένο μας θέμα των αυτοκινήτων. Θα σας παρακαλέσω να θυμηθείτε ε, την συζήτηση για το διοξίδιο του άνθρακα, ότι ο κόσμος χάνεται. Ε, είχαμε ε, συνθήματα, επιχειρήματα και δεν θα πρέπει μόνο να ακούμε τους κατασκευαστές των αυτοκινήτων. Εγώ θα ήθελα να πω αυτό που είπε ο κύριος ε, Ζίπερ. Ε, ο θόρυβος αρρωσταίνει τον κόσμο και εγώ δεν είμαι πολύ ευαίσθητος, ε, αλλά όταν κάποιος συνέχεια ακούει θόρυβο, τότε πραγματικά αυτό είναι πρόβλημα. Και θα πρέπει στα σοβαρά να πάρουμε το θέμα και να το προσεγγίσουμε φιλόδοξα. Αυτό είναι σωστό κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό και και θα ήθελα να ακολουθήσω τον εισηγητή με κάποιε ενδεχόμενες προσαρμογέ. Η γενική κατεύθυνση πάντω είναι σωστή. Και άλλωστε τα πιο ήσυχα αυτοκίνητα ε, μια χαρά απολούνται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μάρτιν Κέλλερμαν. Ενάμιση λεπτό παρακαλώ. Μάρτιν Κέλλερμαν. Δεν κατάλαβα ότι έγινε Ολλανδό ε, από τη μια στιγμή στην άλλη. Εντάξει, ε, θα ήταν ε, όχι τόσο κακό, αλλά όχι για να είναι κανείς να παίζει ποδόσφαιρο. Αλλά ας μην πιάσουμε την κουβέντα τώρα για το Euro. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Μύριο Σλαβιά για την εξαιρετική σκληρή δουλειά που έχει κάνει, γιατί είναι πολύ τεχνικό το ζήτημα Έχω και εγώ ασχοληθεί με τέτοια τεχνικά ζητήματα και ξέρω πόση δουλειά απαιτείται. Τα περισσότερα έχουν καλυφθεί, δεν θα επαναλάβω λοιπόν πράγματα που έχουν υποθεί. Θα ήθελα όμως ε, κάτι πολύ απλό να πω. Δηλαδή ότι φυσικά και στηρίζω τις τροπολογίες ε, του φαινομένου του κυρίου Ούσκη και του κυρίου Ταταρέλα για μια επιπλέον κατηγορία ταξινόμησης ε, για ειδικά οχήματα ειδική χρήση. Η κυρία Μέρκη ε, κάνει λάθο όταν λέει ότι εμεί θέλουμε να εξαιρεθούν τα οχήματα αυτά από την πρόταση. Αυτό είναι ένα σημαντικό επιχείρημα, πρέπει να το διατυπώσουμε. Θέλουμε απλά να υπάρχει μια ξεχωριστή ταξινόμηση, γιατί πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητέ του στην αγορά, να αναγνωριστούν και οι κατασκευαστέ των οχημάτων αυτών, να περιλαμβάνονται στην πρόταση. Οχήματα δηλαδή που παράγονται συνήθω από μικρέ ε, επιχειρήσει, ε, μικρομεσαίε, ω επιτοπλίστων και υπάρχουν εξειδικευμένοι κατασκευαστές σε κάποιες χώρες που έχουν ηγετική θέση στον τομέα αυτό, είναι καινοτόμοι και ε, μιλάμε βέβαια για πολύ μικρές ε, σειρές ε, οχημάτων, βγαίνουν πολύ λίγα μοντέλα, το 0,3% της αγοράς, το πολύ καταλαμβάνουν. Πρέπει να λυθούν υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Μάρτιν, ε, στις ε, ε παρεμβάσεις ε, δεν έχουμε πρόσθετο χρόνο. Ο Ζιλ Περνιό είναι ο επόμενος ομιλητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού εγκρίναμε χθε ε, το δικό μου σχέδιο γνωμοδότηση για τον κανονισμό αυτό που αφορά την ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων. Και μετά από μακρέ διαπραγματεύσει με του κοιόδη συζητητέ και του ε, συντάκτε τροπολογιών, καταλήξαμε σε μια σειρά συμβιβαστικών προτάσεων, ιδίω σε ό,τι αφορά την μνήμα σε μια ολοκληρωμένη συνολική προσέγγιση για τη σημασία που έχει να έχουμε έναν, τον ελάχιστο δυνατό ε, θόρυβο και για τα ηλεκτροκίνητα και υβρεδικά οχήματα. Το πιο δύσκολο ήταν αυτό βέβαια που αφορούσε τις οριακές τιμές του παρακτήματος 3 της πρότασης κανονισμού. Λέω απλά στους συναδέλφους μου από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ότι παρά τις προτάσεις ε, τροπολογιών που ήταν πολύ διαμετρικά αντίθετες πολλές φορές, καταφέραμε εγώ και Σκιώδης από ε, συγκεκριμένα από το ΕΛΚΟ κύριο Κόζα, να καταλήξουμε σε συμβιβαστική ε, τροπολογία που νομίζω ότι μας επιτρέπει να βρούμε την πλέον μετριοπαθή και ισορροπημένη λύση στο μέτρο του δυνατού. Του δυνατού. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις διάφορες προτάσεις που ορισμένες από αυτές επαναλαμβάνουν αυτόματα τις προτάσεις ε, της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ενώ άλλες, άλλες προτάσεις θα μπορούσαν εν τέλει να θέσουν σε κίνδυνο την αυτοκινητοβιομηχανία. Βρήκαμε λοιπόν το συμβιβασμό μεταξύ των δύο αυτών τάσεων. Ο εισηγητής από την Επιτροπή Μεταφορών είπε ότι υπήρξε μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή Μεταφορών χθε που στήριξε τη συμβαστική αυτή πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μάντερ, 1,5 λεπτό παρακαλώ. Το συγγνώμη πριν που πήρα το μικρόφωνο, αλλά κοιτάζατε εμένα κύριε Πρόεδρε και μπερδεύτηκα. Θα ήθελα να επανέλθω αν με επιτρέπετε σε αυτά που είπε ο συνάδελφο Κράμε και κάποιοι άλλοι. Ε, νομίζω ότι έχουμε μεν τις ίδιες προθέσεις, αλλά με διαφορετικό τρόπο θέλουμε να πετύχουμε τον ίδιο στόχο. Νομίζω ότι ο Αντρέας Φαπ ε, πριν από δύο-τρία χρόνια ήταν εισηγητής για τα ελαστικά των ε, οχημάτων και είχαμε έρθει σε επαφή με την ε, βιομηχανία. Η Μισελέν μας είχε πει ότι ναι, συμφωνούμε με πιο δρακόντια μέτρα διότι ο ευρωπαϊκός κλάδος ε, έχει μεγάλο προβάθισμα εναντί των ανταγωνιστών. Και εμείς ε, στοιχηματίζουμε υπέρ της καινοτομίας, μας είχαν πει. Άρα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στον ευρωπαϊκό κλάδο της αυτοκινητομηχανίας να διατηρήσει το προβάδισμα που έχει και να ενθαρρύνουμε ακόμη περισσότερο την καινοτομία, διότι αυτό είναι καλό για την απασχόληση και για την οικονομία όμως. Αν τεθεί σε ισχύ ε, την προβλεπόμενη χρονική στιγμή ο κανονισμός για τα ελαστικά, το 60% των οχημάτων θα μπορούν να ε, τηρήσουν αυτό το όριο, το πρώτο όριο που έχει τεθεί. Και θα μπορεί η μηχανία με την ισχύ της να επεξεργαστεί νέους τύπους οχημάτων που επαναλαμβάνω θα έχουν το προβάδισμα και θα μπορούν έτσι να ανταγωνίσουν αυτά τα οχήματα άλλα οχήματα άλλων κατασκευαστών. Ο Βιτόριο Πρόντι, ευχαριστώ. Νομίζω ότι η εκπομπή θορύβου εξαρτά πολύ από τη χρήση του αυτοκινήτου. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικότερο στα κατοικημένα κέντρα να καθορίσουμε όρια ταχύτητας και υποδομές για να γίνεται σεβαστό το όριο ταχύτητας. Εν γένει ο θόρυβος μετά εξαρτάται και από το αυτοκίνητο και από την οδική υποδομή. Και θα πρέπει εδώ να ενδιαφερθούμε για τα φράγματα κατά του θορύβου, αν θέλουμε να δούμε το όλο σύστημα. Εγώ θα ξεκινούσα από τις μοτοσυκλέτες και τα μοτοποδήλατα, να περιορίσουμε εκεί το θόρυβο, γιατί αυτό στις πόλεις ε, είναι που συμβαίνει. Για τα αυτοκίνητα Προφανώς υπάρχει ιδιαίτερη εκπομπή θορύβου από τον κινητήρα τη στιγμή που ανάβει το πράσινο φανάρι στο σηματοδότη, ξεκινάνε τα αυτοκίνητα και χρησιμοποιούν πολύ γκάζι οι χρήστες. Η μόνη λύση θα μπορούσε να είναι ο περιορισμός της ισχύω ε, τουλάχιστον στα κατοικημένα κέντρα. Ευχαριστώ τον Βιτόριο Πρώτη να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ο κύριος Ζαν θα μιλήσει εκ μέρους της Επιτροπής. Παρακαλώ. Δεν θέλει η Κομισιόν να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τη συζήτηση που ακούσαμε. Το πρώτο στοιχείο αφορά την ολοκληρωμένη ε, προσέγγιση που είναι επιθυμητή. Φυσικά η πρόταση αφορά μόνο τον θόρυβο που εκπέμπουν τα οχήματα και συμπληρώνω την πρόταση για τον θόρυβο από τα ελαστικά που ανέφερε και ο κύριος Μάντερς. Βέβαια και εμείς ε, είμαστε ευαίσθητοι απέναντι στο ότι όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα είναι και πιο συνεκτική ε, στο τεφά τη διατάξη για το θόρυβο. Πριν από λίγες εβδομάδες όλοι οι φορείς, τα κράτη-μέλη, πρόσωποι τη Κομισιόν, εκπρόσωποι ε, οργανώσεων, εκπρόσωποι της βιομηχανίας ε, είχαν ε, συνεδριάσει στο πλαίσιο μιας ομάδας εργασίας για να δουν με ποιο τρόπο μπορεί να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και για το θόρυβο. Και σε ό,τι αφορά την ευθύνη των κρατών μελών επίσης, οι πρόταση που στο τραπέζι Νομίζω ότι πρέπει να ειδωθεί συμπληρωματικά με την έκθεση 1521, ε, την οποία στήριξαν ε, οι 40 συμμετέχοντες, δηλαδή και τα κράτη-μέλη, αλλά και όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Γι' αυτό και εμείς δεν βλέπουμε να υπάρχει αντίφαση μεταξύ της πρότασης αυτής που έχετε μπροστά σας και άλλων μέτρων που θα μπορούσαν να ε, εισαχθούν στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένη προσέγγισης. Δεύτερον, πολλές φορές λέγεται ότι το κείμενο αντικατοπτρίζει τη βούληση να μετρηθεί καλύτερα ε, και η αξία αλλά και η απόδοση των οχημάτων σε ό,τι το θόρυβο. Μέχρι τώρα Κατά το παρελθόν η μέτρηση μετρούσε μόνο την επίδοση του κινητήρα. Αυτό δεν επαρκούσε γιατί όλα τα όρια που είχαν οριστεί δεν μπορούσαν να ορίσουν ακριβώς το θόρυβο όπως να αντιλαμβάνεται ο πολίτης. Θέλαμε λοιπόν να μπορούμε να μετρήσουμε συνολικά το θόρυβο που επέμπει Γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτά τα νέα μέτρα, αυτή η νέα μέτρηση είναι πιο κατάλληλη για να μετρήσουμε ρεαλιστικά ε, τον θόρυβο που, στον οποίο υποβάλλεται ο πολίτης. Με αυτή την μέθοδο επανεξετάζονται λοιπόν οι οριακές τιμές που είχαν οριστεί το 1995 και θέλουμε για κάθε κατηγορία οχήματος, λαμβανομένων υπόψη των του να ορίσουμε κάποιες τιμές συγκεκριμένε. Από ό,τι κατάλαβα θέλουν οι βουλευτές να βάλουν τις προτάσεις τους. Βεβαίως και θα τις εξετάσουμε. Και θα τις δούμε θετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω τέλος το λόγο πάλι στον εισηγητή Πίνο Σλαφούσκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Αυτό το θέμα μας οδήγησε σε πλουσιότατη συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και έχω να πω ένα-δύο πράγματα. Ο κ. Κράμερ είπε ότι το Συμβούλιο περίμενε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περίμενε να μιλήσει πρώτο το Κοινοβούλιο. Και νομίζω γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εμείς θα πρέπει να μειώσουμε το ρυθμό μας. Διότι η τακτική ελιγμή που ακολουθεί το Συμβούλιο δεν είναι σωστή. Δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος θέσπιση νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να μας πιέζουν. Ο Μάρτιν Κάλαναν Ήδη απάντησε στην κυρία Μέρκη. Δεν θέλω εξαιρέσει για τα σπόρα αυτοκίνητα, μόνο ξεχωριστή κατηγορία. Δεν χρειάζεται να πω πολλά για το μακροπρόθεσμο στόχο. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε στόχο. τα δίτροχα και τα τρίτροχα ήδη καλύπτονται. Ε, γνωρίζω ότι θεωρούμε ότι οι μοτοσυκλέτες πράγματι είναι θορυβόδεις. Δεν θα απαγορεύσουμε όμως τις μοτοσυκλέτες και οι νέε μοτοσυκλέτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ΣΥΠΑ ε, καλύπτονται από νομοθεσία. Αν πάει να αγοράσει κανεί μια Harley Davidson σήμερα, ε, η Harley ήδη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις υφιστάμενες προδιαγραφέ. Καλωσορίζω αυτό που ανέφεραν οι συνάδελφοι για τα φορτηγά. 3% των οχημάτων δημιουργούν το 50% του ε, θορύβου. Αυτό τεκμεριώνει τη δική μου θέση, ότι η διαχείριση της κυκλοφορίας και τα όρια ταχύτητας καθώς και οι περιορισμοί κυκλοφορίας των φορτηγών στο κέντρο των πόλεων, όλα αυτά μπορούν να δώσουν πολύ μεγαλύτερα ωφέλη από το να ε, χτυπήσουμε με νέα μέτρα την αυτοκινητοβιομηχανία. Να επενθυμίσω ότι έγινε πριν από κάποια χρόνια. Περάσαμε ένα νόμο για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Όταν το κάναμε αυτό, αυτόματα νομοθετήσαμε για υψηλότερα επίπεδα θορύβου. Γιατί? Διότι ο καλύτερος τρόπος για να μειώσεις τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος είναι να αυξήσεις την απόδοση των κινητήρων. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη παραγωγή θορύβου. Τώρα ζητάμε μείωση επίπεδου θορύβου. Αυτό αυτομάτως το οδηγεί σε μια αύξηση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακο. Και δεν αναπόκειται σε εμά να συζητήσουμε το κόστος που δημιουργεί κάτι τέτοιο στην αυτοκινητοβιομηχανία. Όμως δεν ξέρω αν παρατηρήσατε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία δεν βγάζει μεγάλα κέρδη σε αυτή τη φάση. Η British Leyland, η Jaguar εξαγοράζονται από ειδική ε, εταιρεία. Η Volvo είναι σε κινέζικα χέρια. Δεν ξέρω μέχρι πού θέλετε να φτάσουμε την κουβέντα. Προσβλέπω στις συζητήσεις μας, ελπίζω ότι αυτό που θα πετύχουμε θα είναι η μείωση του θορύβου της κυκλοφορίας προς όφελος της ε, υγείας ε, του, του κόσμου. Ευχαριστώ τον κύριο Μυροσλάφ Ούσκι. Νομίζω ότι ο τομέας των αυτοκινήτων ήδη βρίσκεται σε δυσκολίες και άσχετα από την νομοθεσία αυτή υπάρχουν ε, πολλοί λόγοι γιατί βρισκόμαστε στη θέση αυτή και δεν νομίζω ότι φταίει αναγκαστικά η περιβαλλοντική νομοθεσία. Το θέμα το ανέφεραν αρκετοί. Το θέμα της υγείας και του θορύβου. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με τους συντονιστές, με το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σωστά το θέμα αυτό, διότι όχι μόνο στον τομέα των αυτοκινήτων, αλλά και στους σιδηροδρόμους υπάρχουν σοβαρές συνέπειες ε, για τον πληθυσμό ακόμα περισσότερο δε από, τα, από τους αερολιμένες και αυτό το έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Ε, αλλά μήπως πρέπει να εξετάσουμε την κοινή βάση, ποιες είναι οι συνέπειες ε, για την υγεία από το θόρυβο. Αυτό το συζητήσουμε με τους συντονιστές. Όπως είπε ο εισηγητής, η ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα αναβληθεί στις 19 Σεπτεμβρίου. Το πότε θα πάει το θέμα στην Ολομέλεια θα το δούμε. Ο εισηγητή θέλει να έχει περισσότερε συναντήσει με του σκιώδεις εισηγητέ. Ε, γι' αυτό θέλουμε ευελιξία. Σα ευχαριστώ πολύ. Φτάνουμε στο επόμενο θέμα της ημερησία διάταξη, το υπαριθμόν 4. Σοβαρέ διασυνοριακέ απειλέ για την υγεία. Εδώ ο εισηγητή μα είναι ο Ζιλ Περνιό, Παρνιό και θα ήθελα να του δώσω το λόγο. Παρακαλώ, Ζιλ. Monsieur le Président, chers collègues, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Από τις 11 Μαΐου έχει γνωρίσει αυτό το θέμα ο κύριος Ματίας Γκρότ. Ήθελε να ζητήσει τη γνώμη της νομικής υπηρεσίας όσον αφορά την ακρόση που αφορά την πρότασή μας, την πρόταση της Επιτροπής, όσον αφορά τις διασυνοριακές απειλές που είναι σοβαρές για την ε, υγεία. Μετά την επιστολή αυτό αυτή σαν εισηγητής θέλαμε να, σαν εισηγητές θέλαμε να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή του συστήματος έγκαιρης ε, προειδοποίησης για κάθε σοβαρή απειλή διασυνοριακή για την υγεία. Και ούτω τρόπος θέλουμε να καλύψουμε τα κενά που εντοπίστηκαν τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την κοινοποίηση, την εποπτεία, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων όσον αφορά την υγεία αντίθετα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρώ ότι οι διασυνοριακές απειλές που είναι σοβαρές για την υγεία και οφείλονται στην ιονίζουσα ακτινοβολία θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα της γενικής προσέγγισης που συστήνεται από την παρούσα απόφαση. Το ατύχημα το πυρηνικό του Μαρτίου 2010 στη Φουκουσίμα μας υπενθυμίζει πόσο είναι κρίσιμη σημασία να είμαστε θέση να αντιδρούμε γρήγορα. Λίγη ησυχία λέει ο πρόεδρος παρακαλώ. Γιατί δεν ακούγεται επιτρέψτε του να παρουσιάσει το σχέδιο ε, γνωμοδότησής του, ε, το σχέδιο έκθεσής του και όποιος ε, θέλει να συζητήσει κατά τα άλλα ας ε, καταλήψει την αίθουσα. Το λόγο λοιπόν έχει ο Ζιλ Παρνιό για να μπορέσει ήσυχα να παρουσιάσει την έκθεσή του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να μπορείτε να μου ακούτε και με τα δύο αυτιά άμα γίνει Λοιπόν, θεωρήσαμε αναγκαίο να ζητήσουμε από τι νομικέ υπηρεσίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καθορίσουμε κατά πόσο η νομική βάση τη αποφάσεω θα πρέπει να τροποποιηθεί, αν θα προτείνουμε να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή ε, για ε, πυρηνικό ατύχημα ή ατύχημα που αφορά ραδιενέργεια. Μα διανεμήθη η γνωμοδότηση, είναι πιστευτικού χαρακτήρα Μα δόθηκε στην αρχή τη συνεδριάσεω και η νομική υπηρεσία μα είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη για αλλαγή τη νομική βάσεω τη παρούση προτάσεω. Παρόλο και που στην περίπτωση η δική μα Επιτροπή του Περιβάλλοντο θα ήθελε να διευρύνει το πεδίο εφαρμογή, ούτω ώστε να καλύπτονται και απειλέ που απορρέουν από ε, πυρηνικό ατύχημα ή ακτινοβολία ε, ραδιενέργεια και εφόσον είναι κάτι που απορρέει από την ίδια πρόταση. Και αυτό επιμένω ε, να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή τη παρούσα αποφάση για τι διασυνοριακέ απειλέ που είναι σοβαρέ για την υγεία ε, λόγω ε, ιονίζουσα ακτινοβολία. Αυτό εντάσσεται στη γενική προσέγγιση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει της, του άρθρου 1 της απόφασης. Προς ενημέρωσή σας, υπέβαλα σήμερα την έκθεσή μου στην υπηρεσία μετάφρασης. Θα γίνει μια παρουσίαση λεπτομερής στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, στις 10 Ιουλίου ε, και η προθεσμία ε, υποβολής τροπολογιών έχει καθοριστεί 18 Ιουλίου. Σε αυτό το στάδιο θέτηση τη ε, εκθέσεω στην Επιτροπή Περιβάλλοντο προβλέπεται, κύριε Πρόεδρε, για τι 18 Σεπτεμβρίου, ενώ ψηφοθέτηση στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πολύ τον Ζιλ Παρνιό. Οι σκιώδεις εισηγητές έχουν το λόγο. Ο Κρίστοφερ Φιέλνερ. Ε, διάβασα την έκθεση της νομικής υπηρεσίας. Νομίζω ότι είναι αρκετά λογική και δεν δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε τι έχει να μας πει η νομική υπηρεσία. Καμιά φορά μας λένε κάποια πράγματα που δεν έχουν υποβάλει γραπτός. Λοιπόν, θα θέλαμε να ακούσουμε τα σχόλια της νομικής υπηρεσίας σχετικά με την ομοδότησή της. Ευχαριστώ, συνάδελφος Ρεμπέκα Τέιλορ. Um, um, να πω ότι διάβασα την ε, νομική άποψη και δεν έχω ανησυχίες ε, ούτε εγώ, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε τα σχόλια της ε, νομικής υπηρεσίας. Η Φρίντα Ρίποτς, σκιώδης εισηγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στα πλαίσια της νομικής αυτής συμβουλής που μας δόθηκε, θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι είναι ευπρόσδεκτη αυτή η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας που λέει ότι δεν χρειάζεται αλλαγή της νομικής βάσης ακόμα και αν αποφασίσουμε σε Επιτροπή να καλύψουμε και κινδύνους για την υγεία που προκύπτουν από ιονίζουσα ακτινοβολία. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό, διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαμε μέχρι τώρα υπήρξαν κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την εξαίρεση της ιονίζουσης ακτινοβολίας και θα ήθελα να ζητήσω να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσο όλες οι συνέπειες για τη δημόσια υγεία από πλευρά ιονίζουσας ακτινοβολίας καλύπτονται από τη συνθήκη Euratom διότι φαίνεται να υπάρχουν κάποιες ε, αμφιβολίες και δοθέτων των στόχων της Πρωτές Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήταν λογικότερο να καλύπτονται κίνδυνοι για την υγεία που απορρέουν από την ιονίζουσα ακτινοβολία σε αυτή την πρόταση και χαίρομαι που ο εισηγητής ε, το πρότεινε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για το ECR, ο Μίλαν Κάμπτοχ. Εδώ ήτανε. Μόλις τον είδα. Από ό,τι δεν βλέπω δεν είναι εδώ. Προχωράμε λοιπόν. Γύριμα στα λάκα. Επίσης δεν είναι εδώ. Ο κύριος Κυλακάκης επίσης δεν είναι παρόν. Ωραία. Η κυρία Κούκοβιτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προφανώς οι διασυνοριακές απειλές για την υγεία είναι τόσο απομακρές τόσο μικρή αυτή η κίνδυνη που είναι σοβαρό πρόβλημα, αλλά δεν είμαστε πολύ παρότι συζητήσουμε το θέμα. Αυτό δείχνει πόσο χαμηλή είναι η ευαισθητοποίηση για αυτά τα προβλήματα. Ε, είναι χαμηλή ευαισθητοποίηση και εντό ε, Ευρώπης και πέρα από τα σύνορα. Διότι τα προβλήματα που μπορούν να διοργηθούν, τα διασυνοριακά, μπορούν να επηρεάσουν την υγεία ανθρώπων και να πλήξουν και την οικονομία. Πρέπει να δούμε ποιε είναι οι συνέπειε του προβλήματο αυτού όσον αφορά και τα εθνικά εισοδήματα, από πλευρά οικονομική δηλαδή. Και για την κοινωνία που θέλει να επιβιώσει. Είδαμε τι είχε γίνει παλιά και στην Κίνα με την γρήπη των πτηνών. Το 2008 όταν η Σλοβενία είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβληματιζόταν γιατί τι θα έπρεπε να κάνει να συμβεί κάτι παρόμοιο. Ετοιμότητα λοιπόν. Η ετοιμότητα είναι ύψης της σημασίας. Γι' αυτό υποστηρίζω την προσέγγιση που ακολουθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει κύριε Ριβάζη. Να επανέλθουμε στην ουσία. Είναι σημαντικό ζήτημα. Να σας δώσω δύο παραδείγματα που δείχνουν ότι θα πρέπει να έχουμε πληροφορίες και είναι σημαντικό αυτό. Είχαμε το τύχημα της Φουκουσίμα. Ο κύριος Παρνιώτα ανέφερε και είχε, είχαμε σημαντικό ατύχημα το 2011. Είχαμε την ενεργό σύννεφο με ιόδιο που διέτρεξε όλη την Ευρώπη επί ένα μήνα και δεν γνωρίζαμε από πού δημιουργήθηκε την προέλευση. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Με ένα μήνα μετά είδαμε ότι ήταν από την Ουγγαρία, από ένα Ινστιτούτο που παρήγαγε ε, ραδιενεργές ε, πηγές, υλικό που περιείχε ιόδιο. Ποιες είναι οι πληροφορίες ότι στα κράτη-μέλη δεν υπήρχαν μέσα μέτρηση της ραδιενέργειας. Ακτινοβολία και μέσω ενεργού άνθρακα που θα μπορούσε να εντοπίσει τα ραδιενεργά αέρια. Είχαν ραδιομέτρα μέτρηση ραδιενέργειας μόνο απλά τα κράτη-μέλη. Να επιθυμίσω κάτι στο Ζιλ Παχνιό. Σύμφωνα με τη συνθήκη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων υπάρχουν χώρες όπως η Σουηδία και η Γερμανία, δύο χώρες που έχουν σα, σαφή μέτρα για τη ραδιενέργεια αλλά έχουν δικαίωμα να κοινοποιούν στο κοινό τα μέτρα. Αυτό είναι στα πλαίσια της συνθήκης για τη μη διάδοση. Πρέπει να πούμε ότι αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να είναι δημόσια γιατί αυτοί που ήταν κοντά σε αυτό το Ινστιτούτο στην Ουγγαρία δεν ξέρουμε σε τι δόσεις εξετέθησαν. Θέλουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε έκθεση τι δόσεις ε, έχουν υποστεί ραδιενέργειες οι άνθρωποι που είναι κοντά σε αυτό το Ινστιτούτο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα ε, διασυνολογικού χαρακτήρα που πλήττει τον κόσμο. Η, Ντάγμα Ευχαριστώ πολύ. Διάβασα και εγώ τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας και όπως πάντα είναι εξαιρετική ε, και δεν είναι καθόλου λάθος, αλλά αυτό που θα επιθυμούσα εγώ από τη νομική υπηρεσία μας, και το ξέρουν ε, αυτό οι συνάδελφοι, θα ήθελα η νομική υπηρεσία να λαμβάνει υπόψη ότι είμαστε πολιτικό θεσμικό όργανο. Και ως νομικός εγώ θα ήθελα να παρουσιάζουν μεν την νομική ε, κατάσταση, αλλά να παρουσιάζουν και τη δυνατότητα να πετύχουμε έναν πολιτικό στόχο. Ο πολιτικός στόχος εδώ είναι στην έκθεση να υποδεικνύουμε ότι υπάρχει σοβαρή διασυνορική απειλή για την υγεία μέσω της ε, ε, τη πυρηνική ακτινοβολία. Και ξέρουμε ότι αυτό καλύπτεται από τη συνθήκη Euratom, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Στην έκθεση αυτή θέλουμε να το τονίσουμε και όχι μετά από κάποιο ενδεχόμενο ατύχημα. Υπάρχουν διάφορες απειλές ε, από πυρηνικά απόβλητα, ακτινοβολία. Ξέρετε ότι υπήρξαν και ε, απειλές κατά προσώπων ε, με πυρηνικά μέσα και σε μια τέτοια έκθεση είναι καλό να το αναφέρουμε αυτό Φυσικά το θέμα της ε, Ιωνίου Ακτινοβολία καλύπτεται από τη συνθήκη Euratom, αλλά εγώ νομίζω ότι πολιτικά είναι απαραίτητο να το ε, επαναλάβουμε και μπορούμε ως κοινοβουλίο να το κάνουμε αυτό. Και γνωρίζουμε φυσικά τις διάφορε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο παρελθόν όμως. Έχουμε επιλέξει τις νομικές βάσεις που θέλαμε από πολιτικής πλευράς. Αυτό δεν είναι πολύ καθαρό πάντα από νομικής πλευράς και καταλαβαίνω τους συναδέλφους από την νομική υπηρεσία που δεν μπορούν να το εγκρίνουν αυτό νομικά. Πολιτικά όμως συχνά πρόκειται για μια δήλωση και γι' αυτό θέλω πολιτικά να αποφασίζουμε ποια νομική βάση θέλουμε. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Μετά μπορούμε να διαπραγματευτούμε και με την Κομισιόν και στο παρελθόν είχαμε επιτυχία. Ξέρετε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανειλημμένα έχει πει «Ωραία, συμφωνήσουμε και με τη δεύτερη νομική βάση». Ω προ το περιεχόμενο, δεν, θα, θέλω καθόλου να το ξελογήσω αυτό. Αυτό θα το κάνει ο εισηγητή με του σκιώδει. Αλλά θα ήθελα να σα προειδοποιήσω, εάν θέλουμε να κάνουμε μια πολιτική δήλωση, κάτι που βρίσκω σωστό, ε, να συμπεριλάβουμε και τον κίνδυνο από ε, ε, την πυρηνική ακτινοβολία και να μην το αποφύγουμε. Και γι' αυτό με όλο το σεβασμό προς τους συναδέρφους από την νομική υπηρεσία παρακαλώ να μεταφέρετε και στον κύριο Τρέξλερ που συνυπέγραψε την γνωμοδότηση. Θα ήθελα στην γνωμοδότηση την ε, νομική θέση, αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν για να πετύχουμε έναν πολιτικό στόχο. Ευχαριστώ πολύ, ο Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συνεχίσω πάνω στην παρατήρηση του συναδέλφου Ζιλ Μπαχνιού για να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι να εξετάσουμε τις ιονίζουσες ακτινοβολίες που μπορούν ε, να μεταφερθούν από μετεωρολογικά φαινόμενα και μέσω τροφίμων που εισάγονται στην Ευρώπη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω πως κάποιες πτυχές όπως του μαύρου άνθρακα, black carbon, της εθάλης, έχει σημασία και για την θέρμανση του πλανήτη και δημιουργεί ανησυχίες για την υγεία, διότι πρόκειται περί σωματιδίων που μπορούν να εμπεριέχουν καρκινογόνες ουσίες. Υπάρχει ένα σύνολο πραγμάτων που πολλών που πρέπει να λαμβάνονται όσοι πτυχές υπόψη χωρίς να λησμονούμε καμία. Ευχαριστώ κύριε Πρώτη. Ευχαριστώ και καθότι είναι εδώ η νομική υπηρεσία να δώσω τον λόγο στον κύριο Ροτρίγκες που εκπροσωπεί τη νομική υπηρεσία διότι αναφέρθηκε επανειλημμένη γνωμοδότηση. Σας παρακαλώ κύριε Ροτρίγκες. Uh, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω σε αυτά που γράψαμε στην ε, γνωμοδότησή μας της νομικής υπηρεσίας μόνο που ετέθη το θέμα να γνωρίζουμε κατά πόσο η συμπερίληψη ιονίζουσας ακτινοβολίας που προέρχεται από ατυχήματα θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το νομοθέτημα. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο, κατά πόσο η νομική βάση θα έπρεπε να αλλάξει. Ήταν νομικό ερώτημα που απευθυνόταν από νομική υπηρεσία που έδωσε νομική γνωμοδότηση. Η νομική γνωμοδότηση συνεπέρανε ότι βλέποντας το στόχο και το περιεχόμενο της πρότασης που είναι βασικός προσανατολισμός που πρέπει να ακολουθήσουμε για την αξιολόγηση της νομικής βάσης, έχοντας δει λοιπόν το περιεχόμενο και την εμβέλεια της προτάσεως, είναι δυνατόν να παραμείνει η παρούσα νομική βάση για τη δημόσια υγεία που εδράζεται τη συνθήκη σε λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και δεν χρειάζεται να προσθεθεί η νομική βάση του άρθρου 32 της συνθήκης Ευρατών. Η νομική λογική που ακολουθήσαμε κατέληγε στο ότι βασικός στόχος, ο κύριος στόχος της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υποστήριξη πολύ στο άθρο ένα, την πρόληψη και τον έλεγχο σοβαρών ανθρωπίνων ασθενειών σε όλα τα κράτη-μέλη και να εξαλειφθούν με σημαντικές πηγές διασυνοριακών απειλών. Λαμβάνοντας υπόψη το στόχο και το γενικό περιεχόμενο της προτάσεως, είναι σαφές ότι ο βασικός στόχος πρέπει να δικαιολογεί τη νομική βάση. Και η σωστή νομική βάση πρέπει να είναι η βάση για την δημόσια υγεία, ως έχει δηλαδή το ότι μία απειλή μπορεί να δημιουργείται από ιονίζουσα ακτινοβολία, αυτό δεν απαιτεί απαραίτητα διάταξη της συνθήκης Ευρατόμου να προσθεθεί στη νομική βάση. Το συμπεράναμε αυτό βάσει της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που λέει βασικά ότι όταν υπάρχουν δύο βασικοί στόχοι ή δύο στόχοι, τότε ο βασικός, ο κεντρικός στόχος επικρατεί. Και εδώ κεντρικός στόχος είναι η αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών για τη υγεία και το γεγονός ότι μία από τις απειλές ίσως να προέρχεται από ραδιενεργή πηγή δεν απαιτεί προσθήκη νομικής βάσης της Ευρατόμ. Να προβώ ένα τελευταίο σχόλιο. Αυτό το δικό μας συμπέρασμα βάσει της επιστολής που μας αποστήλατε και λαμβάνω δεόντως υπόψη της παρατήρησης της κυρίας Ροτ Μπέρεντ, τις οποίες καταλαβαίνω, όπως σας είπα, ο ρόλος μας ως νομική υπηρεσία πάντα εδράζεται επί του αιτήματο της επιστολής. Και αυτό κάναμε χρησιμοποιώντας νομική προσέγγιση επιχειρηματολογία βέβαια. Πρακτικό ερώτημα όμως τώρα. Αν η Επιτροπή σας αποφασίσει να παρουσιάσει, να υποβάλει τροπολογίες ή αν επιθυμούσε να κάνει κάτι τέτοιο για να προσθεθεί η νομική βάση της Ευρατόμ, που δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο από τη συζήτηση, τότε η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θα πρέπει να τοποθετηθεί και να γνωμοδοτήσει. Εφόσον συμπεράναμε ότι δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο και από ό,τι είδα από τη συζήτηση όλοι συμφωνούν, νομίζω ότι η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη. Άρα είναι δυνατόν να παραμείνει η ισχύουσα νομική βάση. Ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχει άλλη ερώτηση, με τα χαράς να απαντήσω. Ευχαριστώ κύριε Ροτρίκες, ε, αλλά τώρα έχουμε δύο ακόμα ε, παρεμβάσεις, η κυρία Ροτμπέρεντ και μετά ο κύριος ε, Παρνιό. Δύο ερωτήσεις. Δύο, δύο ερωτήσεις. Η πρώτη, σε ό,τι αφορά την νομική γνωμοδότηση. Πρώτο ερώτημα. Εάν προσθέταμε σοβαρές δυσνορικές απειλές ε, λόγω ατυχήματος ή ραδιενέργειας. Πιστεύετε ότι αυτό είναι δευτερεύον στην πρόταση. Εγώ νομίζω ότι πρόκειται για ανεξάρτητη απειλή και ανεξάρτητο κίνδυνο. Το δεύτερο ερώτημα νομικό. Αν αφήσουμε ως δευτερεύουσα βάση νομική την Ευρατόμ, αλλά θέσουμε ζήτημα σοβαρή απειλή απειλή ή οντίστοιχη ακτινοβολία. Η τη ακτινοβολια η κομισιον το Συμβούλιο ή άλλοι νομομαθεί μπορούν να μα πούν ότι δεν μπορεί να μπει γιατί καλύπτεται από την συνθήκη Ευρατών. Ευχαριστώ, ο Ζήλ Παρνιό. Euh, Είναι πολύ ενδιαφέρον ε, και ε, γενικά όλο αυτό που συζητήσαμε, αλλά και ανταλλαγή απόψεων με την Dagmar. Ουσιαστικά έχουμε αυτή την νομοθεσία, θέλουμε να εκπονήσουμε μια απόφαση για τις σοβαρές διασυνορικές απειλές για την υγεία και η πρώτη επαφή που είχα ως εισηγητής με τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν θέλησα από πολιτική πλευρά, γιατί θεωρώ ότι είναι από πολιτική πλευρά σημαντικό, να διευρύνουμε, να επεκτείνουμε όλα τα σχετικά με την ραδιενέργεια, την οντίζουσα ακτινοβολία, σε αυτήν την πολιτική απόφαση, μου είπαν ευθύ εξ αρχή αδύνατον. Αδύνατον γιατί έχουμε τη συνθήκη βρατό. Από πολιτική πλευρά λοιπόν δεν μπορείτε να τροποποιήσετε εσεί το αντικείμενο. Μα ξέρετε κι εγώ νομομαθή είμαι. Δεν είμαι μόνο βουλευτή, είμαι νομικός και μέσω του αγαπητού Προέδρου, είπα θα ζητήσω τη νομική γνωμοδότηση από τη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, που μου λέει πλέον στη νομική της γνωμοδότηση ότι ο αρχικός μου πολιτικός στόχος, δηλαδή να ενσωματώσω όλα τα στοιχεία, δηλαδή ενέργεια, ακτινοβολία, η ενσωμάτωση όλων αυτών λοιπόν, και θα το συστήσουμε επί της ουσίας στις ε, 18 Ιουλίου, μου το επιτρέπει, εξού και χαίρομαι πάρα πολύ που είχαμε αυτή τη νομική γνωμοδότηση και χαίρομαι και ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο που απέστειλε την επιστολή αυτή στις 11 Μαΐου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν εμείς πολιτικά να εργαζόμαστε λαμβάνοντας υπόψη την νομική γνωμοδότηση ώστε να έχουμε μια απόφαση η οποία κατά την άποψή μου τουλάχιστον θα βελτιωθεί γιατί θα μπορεί να λάβει υπόψη το σύνολο των διασυνοριακών απειλών σαν αυτές που έχουμε ήδη βιώσει και σαν αυτές που μας ανέφερε, παράδειγμα χάρη με το παράδειγμα του συγκεκριμένου, η συνάδελφος Μισελ Ριβαζή. Σημαντικό πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα που δεν περιορίστηκε στο έδαφος ε, της Ουγγαρίας το 2011 και ήταν ένα θέμα το οποίο διακύβευσε και την υγεία των συμπολιτών μας. Rodriguez, würden Sie das Κύριε Ρωτρίκη, θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, πολύ σύντομα να απαντήσω στα δύο ερωτήματα. Να ευχαριστήσω την κυρία Ροτμπέρεν που τα έθεσε. Είναι δυνατό να προστίθενται κανόνες διατάξεις για, σε σχέση με ατυχήματα τα οποία προέρχονται, οφείλονται σε ραδιενέργεια ή κάποιο άλλο ε, έκτακτο ε, περιστατικό. θα πρέπει να συμπεριληφθεί μια νέα δέσμη μέτρων σε αυτή την περίπτωση. Και έχουμε μια απόφαση ε, του Συμβουλίου από το 87 για πρόορια ανταλλαγή δεδομένων σε περίπτωση ε, έκτακτης ανάγκης λόγω ρεδινές. Αυτός πρέπει να, αυτές οι διατάξεις πρέπει να ακυρωθούν, να καταργηθούν, αν υπάρξει αυτή η νέα ε, απόφαση. Αντικαθίσταται δηλαδή το νέο σύστημα και έχουμε ένα νέο γενικό σύστημα που καλύπτει και την ανταλλαγή πληροφοριών που απαιτείται για την αντιμετώπιση αυτής της σοβαρής διασυνοριακής απειλής που προέρχεται από ένα έκτακτο περιστατικό με ραδιενέργεια. Στο σημείο 15 επίσης λέμε ότι αν το Συμβούλιο, όπως πολύ σωστά πείτε Συμβούλιο ή Κομισιόν, ίσω και κατά πάσα πιθανότητα θα το κάνουν, ίσω έρθει και πούνε ότι θέλουμε τη νομική βάση τη Ευρατόμ που ήδη υπάρχει. Αυτή τη στιγμή κρεμεί μια υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια διαφορά για την καταλληλότητα ή μη μια συνδυασμένη νομική βάση μεταξύ τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη Ευρατόμ. Και εμεί υποστηρίζουμε ότι η νομική βάση θα πρέπει να είναι μόνο η ενέργεια. Άρα συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν χρειάζεται ε, νομική βάση ευρατών. Έχουμε μόνο την γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα μέχρι στιγμή. Αυτό μας δίνει βέβαια πάντα κάποια ένδειξη. Αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, και για να είμαι σύντομο, θα σα πω πολύ απλά ότι αφορά η υπόθεση έναν κανονισμό για κοινοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακέ υποδομέ. Λοιπόν, η Κομισιόν και το Συμβούλιο θεωρούν ότι το γεγονό ότι υπάρχει αναφορά σε επενδύσει στο τομέα της ενέργειας από μεταδενεργές πηγές, το γεγονός ότι ο κανονισμός περιλαμβάνει αυτή την έδειξη, αυτή τη διάταξη, ε, σημαίνει ότι απαιτείται η νομική βάση ευρατών. Εμεί ε, δεν συμφωνούμε και προσβάλαμε αυτή την απόφαση στο δικαστήριο. Εμείς πιστεύουμε ότι η νομική βάση για την ενέργεια, δυνάμει της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί. Και βέβαια τώρα πρέπει να περιμένουμε την τελική ετοιμιγορία του δικαστηρίου. Όλα αυτά τα λέω για να σας πω ουσιαστικά ότι γνωρίζουμε ότι αν συμπεριλάβουμε τις νέες αυτές απειλές που προκύπτουν από κάποιο συμβάν που έχει να κάνει με ραδιενέργεια, θα πρέπει να ακυρωθεί η νομοθεσία του 87 που αφορά μόνο αυτό το πράγμα και θα πρέπει στο κείμενο της πρότασης να αναφέρεται ξεκάθαρα ότι το πρώτο που θέλουμε είναι να ορίσουμε τους μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών κτλ. για να αντιμετωπιστούν ακριβώς αυτές οι σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία. Στο σημείο 10 ε, αναφέρουμε και ένα παράδειγμα του μέσου σταθερότητα κανονισμός το 2006 Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, βάσει άρθρων της συνθήκης για την ε, λειτουργία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον εν κανονισμό έχουμε λίγο πολύ την ίδια δομή όπως και σε αυτή την περίπτωση. Και ο στόχος είναι ο ίδιος. Έχουμε διατάξεις σε ό,τι αφορά ενέργειες με τρίτες χώρες για την εντόπιση σοβαρών απειλών. πριν και μετά την διενέργεια ενό ατυχήματο. Μέτρα που αφορούν την ετοιμότητα, το σχεδιασμό, τη μόνιμη επιτήρηση και εποπτεία, παρακολούθηση, έγκαιρη προειδοποίηση κτλ. Άρα και αυτό είναι ένα μέσο, ένας μηχανισμός που θα μπορούσε να συγκριθεί με το προκείμενο εδώ. Έξω και λέω ότι δεν χρειαζόμαστε την νομική βάση της Ευρατόμ. Ακόμη και αν υπήρχε ανάγκη. Μπορεί, ίσως, να μας, θα μπορούσε να μας βοηθήσει ίσως η απόφαση του δικαστήριου ότι ο βασικός στόχος είναι αυτός εδώ. Υπάρχει και ένα τμήμα που αφορά τη ραδιενέργεια, αλλά δεν σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να προστίθεται η νομική βάση για την Ευρατόμ. Το θέμα είναι ποιο είναι ο βασικό στόχο. Αυτό μετράει. Πάντα αυτό λέει και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και γι' αυτό καταλήξαμε και εμεί στην γνωμοδότησή μα αυτό το συμπέρασμα. Yeah, σας ευχαριστώ πολύ. Ίσως ε, να παραπέμψουμε το θέμα στον κύκλο των σχεδόν εισηγητών να συνεχίσει να συζητιέται εκεί το θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πλήρη ε, γνωμοδότηση και για την ε, επεξήγηση των ερωτημάτων. Το θέμα είναι αν είναι πολιτικά τα θέματα που τίθενται διότι για τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές το θέμα είναι τι είναι πολιτικά εφικτό. Σας ευχαριστώ πάντως θερμά για την γνωμοδότησή σας και την αναλυτική απάντηση. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Η πρόταση εδράζεται επί του άρθρου 168 της συνθήκης που συμπεριλαμβάνει τώρα και αναφορά σε σοβαρέ διασυνοριακέ απειλέ για την υγεία. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι ήταν σημαντικό να επεκταθεί η φυστάμενη νομοθεσία για τι μεταδοτικέ ασθένειε που δεσπίστηκε από το 98 και λειτουργεί καλά για να καλύψουμε και άλλα είδη απειλών από χημικού κινδύνου, ε, περιβαλλοντικέ πηγέ κλπ. Στην τελική σκέψη 7 τη Πρωτεύουσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρητά αναφέρουμε ότι η απόφαση δεν ισχύει για σοβαρές δυσονορικές απειλές για την υγεία που προκύπτουν από ιονίζουσα ακτινοβολία, καθώς αυτές οι απειλές ήδη καλύπτονται από το άρθρο 2 και κεφάλαιο 3 της συνθήκης που ιδρύει την Ευρατόμ. Ήδη λοιπόν υπάρχουν διατάξεις συνθήκης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τις απειλές που προκύπτουν από την ιονίζουσα ακτινοβολία. Γι' αυτό το πεδίο εφαρμογής της προτάσεως Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σαφές. Καλύπτει όλες, όλες σοβαρές δυσυνοριακές απειλές για την υγεία με εξαίρεση αυτές που προκύπτουν από ενίζουσα ακτινοβολία. Η υπόλοιπη πρόταση δεν έχει αναφερθεί σήμερα. Καλύπτει επί παραδείγματι ενίσχυση σχεδιασμού ετοιμότητας, σαν κομμάτι του σχεδιασμού ετοιμότητας. Η εισαγωγή προβλέπεται ε, για την κοινή προμήθεια ε, εμβολίων που ήταν αντίδραση της επιδημίας του 2009. Είχαν αγοράσει οι χώρες τα εμβόλια ξεχωριστά και ήταν διαφορετικές οι συμβάσει. Προτείνουμε λοιπόν μια κοινή, α, κοινό εφοδιασμό όσον αφορά τα εμβόλια. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι δεν εστιάζεται απόλυτα στην ιονίζουσα ακτινοβολία και μόνο το κείμενο. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά κόμματα του κειμένου. Προτείνουμε να χρησιμοποιείται το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ταπόκρισης, αυτό που υπάρχει τώρα σαν μηχανισμός διαβίβασης ε, ε, προειδοποίησεων μεταξύ κρατών μελών και προτείνουμε να χρησιμοποιείται ένα κοινή αξιολόγηση κινδύνων και να χρησιμοποιείται και Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας που είναι η παρούσα επιτροπή που χρησιμοποιείται για το συντονισμό τη ανταπόκριση των κρατών μέλων. Θα ήθελα επίση να πιστήσω την προσοχή και στο άρθρο 12 τη πρόταση που είναι νέο και ενισχύει τις κοινοτικέ διατάξεις που επιτρέπει σαν δίκτυα ασφαλείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω κατεξοδότηση πράξεων να λαμβάνει μέτρα αν κατεπίγους ανάγκη ξεφύγει από τον ένα έχω ξεχωριστού κάτους μέλους. Αυτή είναι μια νέα διάταξη. Επίσης έχουμε εισάγει νέα διάταξη σχετικά με τη διεθνή συνεργασία διότι θεωρούμε ότι αυτού του είδους οι απειλές πολύ συχνά προέρχονται εκτό Ευρωπαϊκή Ενώσεως, αλλά είναι το να έχουμε μια τέτοια διάταξη. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα που συζητήθηκε εκτενώς σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκτιμούσε αν ελάμβανε ένα αντίγραφο τη νομοδοτή νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου σε κάποια φάση τη διαδικασία, ώστε να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε μαζί σα επί του θέματο. Αλλά σίγουρα σε επόμενε συνεδριάσει με τα χαρά να φέρουμε του συναδέλφου που είναι υπεύθυνοι για την Ευρατόμ και για θέματα ευρατόμ, να έρθουν και αυτοί για να μπορέσουν να εξηγήσουν τα σχετικά μέτρα. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ πολύ την Κομισιόν. Ξέρω ότι βρίσκεστε στη μέση και ξέρω επίσης ότι ο ενθουσιασμός ε, στο Συμβούλιο για αυτό το νομοθέτημα είναι κάπως περιορισμένος. Ίσως θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τον ενθουσιασμό αν κάνουμε καλή δουλειά. Τέλος, ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Ζιλ Παρνιό. Παρακαλώ. <coughs> Εντάχει, κύριε Πρόεδρε, έχοντας ακούσει όλες τις παρεμβάσεις των συναδέλφων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Διευθύνσεως της Αρμόδιας, από αυτά που ακούσαμε μόλις τώρα, ίσως μπορώ να προβώ σε κάποια σχόλια όσον αφορά το πλαίσιο της απόφασης που είναι προφανώς πολιτικής χρειάς, όπως τόνισε και συνάδελφος Dagmar Rodberend προηγουμένως. Μέσω της προτάσεως, αποφάσεως, έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τα μαθήματα από διάφορες κρίσεις που αντιμετωπίσουν τελευταία χρόνια. Όπως η επιδημία της ε, γρήπης των πτηνών, το 2009 και το νέφος του ηφαιστείου του 2010 ή το βακτηρίδιο E. coli το 2011 όλη αυτή την περίοδο τα αντιμετωπίσαμε αυτά. Ήταν αναποτελεσματική η προστασία των Ευρωπαίων ανδρών και γυναικών. Άρα χρειάστηκε αυτή η πρόταση που κατέφθασε στις 8 περασμένου Δεκεμβρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσωπικά δέχομαι μεταθέρμης αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή την απόφαση, αυτή που θα συζητήσουμε στις 10 του Ιουλίου, διότι θεωρώ ότι ε, ε, εν μέρη καλύπτει κάποιες ανησυχίες μας, διότι θα πρέπει να επιτρέψουμε μια επέκταση των μέτρων αξιολογήσεων του κινδύνου και να ενισχύσουμε επίσης το ρόλο της Επιτροπής ε, Ασφάλειας και Υγείας και να ετοιμάσουμε καλύτερα ακόμα την καταπολέμηση αυτών των κρίσεων και μετά μας επιτρέπεται και ε, ανάντι και κατάντι να έχουμε κάποιες διατάξεις που προτείνονται. Και θα ήθελα ταυτόχρονα, όπως θα δείτε κατά την έκθεση που θα σας αποσταλεί, θέλω έλεγα διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της απόφασης να καλύπτεται και άλλες απειλές όπως αυτή πέραν αυτών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως ιονίζουσα ακτινοβολία ή ε, τα διάφορα εξοπλισμό ραδιενεργό και έδειξαν και πρόσφατα ε, επεισόδια ότι δεν είναι έτοιμη η τα διαφορα εξοπλισμο ραδιενεργο και εδειξαν και προσφατα Ένωση για να αντιμετωπίσει ε, χάρη ελαττωματικά μηχανήματα ιατρικά και φάρμακα που δεν είναι καλά. Αυτά είναι ευαίσθητα θέματα, όχι μόνο για την κοινή γνώμη, αλλά και για μας. Και πρέπει να κινηθούμε και μέσω του μηχανισμού επιτροπολογή που υφίσαμε πρόσφατα. Άρα το πεδίο εφαρμογή τη παρούσα αποφάση θα πρέπει να διευρυθεί και να καλύπτει τι απειλέ τη λαθασμένη χρήση των φαρμάκων και τη χρήση ε, ε, ε, ελαττωματικών ιατρικών μηχανημάτων. Αυτό ήταν και πρόσφατα στην επικαιρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω και προτάσεις και για τη δημιουργία συντονισμένου μηχανισμού ανταλλαγής ε, κοινοποίησεων. Είχαμε προβλήματα τελευταία χρόνια όσον αφορά και τις εμπειρογνώμονες. Θα πρέπει να επανέλθουμε Προστασία των στοιχείων των προσωπικών επίσης κάτι πρέπει να εξεταστεί. Καλύτερος ορισμός του, της εντολής του Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Ασθενειών. Να επιθυμήσουμε πόσο σημαντική είναι η ενισχυμένη συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις ίδιες χώρες. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και πολύ και μετά θέλουμε να διευκολύνουμε και τις κοινέ διαδικασίες για τα αντίμετρα, τα ιατρικά που πρέπει να εφαρμόζονται και τέλος να υπάρχει τακτικός διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι θεωρώ ότι στον όλο μηχανισμό αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρα από την νομοθετική δουλειά έχει θέση που πρέπει να έχει το διάλογο που χρειάζεται στον αφορά τους κινδύνους θέση. Λοιπόν, με θέρμη και αποφασιστικότητα συντάσσω την έκθεση. Νομίζω ότι έχουμε ένα κείμενο εδώ, θεμελιώδες, για τα 500 εκατομμύρια πολίτες μας, για τα επόμενα χρόνια, κυρίως έναντιον αυτών των κρίσεων που δυστυχώς θα δημιουργηθούν και τα επόμενα χρόνια. Από εμά εξαρτάται όχι μόνο να είμαστε δραστήριοι, αλλά ε, να θεσπίζουμε νομοθεσία που θα προστατεύει καλύτερα εκείνους οι οποίοι μας εκλέγουν, δηλαδή τους Ευρωπαίους άνδρες και γυναίκες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παρνιό. Στις 10 ε, Ιουλίου θα ξαναξετάσουμε την έκθεση εδώ στην Επιτροπή μας ε, και η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 18 Ιουλίου. Ψηφοφορία θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου. Και προβλέπετε να συζητηθεί το θέμα και να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Φτάνουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης ε, που είναι το, τα σημεία 5 και 6. Έχουμε το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία ορίζον 2020. Και έχουμε το ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης για την έρευνα και την καινοτομία. Έχουμε λοιπόν τα θέματα 5 και 6 στην ημερήσια διάταξη. Πολύ σύντομα, παρακαλώ ποιον θέλει να εγκαταλείψει την αίθουσα τώρα, έχει την ευκαιρία για να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το θέμα. Ε, αρμόδια επί της ουσίας είναι η Επιτροπή ε, Βιομηχανίας και θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον ε, εισηγητή Μπουσόη. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, και εγώ ήθελα να σας προτείνω να συζητήσουμε μαζί τα δύο θέματα αυτά, διότι ακολουθούν λίγο πολύ την ίδια γραμμή. Οι δύο προτάσεις που συζητάμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικές για το μέλλον ε, της έρευνας ε, και της καινοτομίας και, εδώ και σε άλλες επιτροπές έχουμε ε, πει ότι χρειαζόμαστε περισσότερη καινοτομία. Η έλλειψη καινοτομίας ε, ήταν ε, μεγάλο μειονέκτημα της Ευρώπης όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Εγώ θέλω να στηρίξω την αριστεία στην επιστήμη και τη σχέση ανάμεσα στην έρευνα και την καινοτομία που θα βοηθήσει την βιομηχανία μας να ανταποκριθεί σε προκλήσεις της κοινωνίας. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των διαφόρων ενδιαφερομένων όπως είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ε, της κοινωνίας. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την σκληρή δουλειά της πάνω στις προτάσεις αυτές. Οι προτάσεις είναι εκθενείς και πιστεύω ότι ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Οι ε, τροπολογίες που προτείνω είναι απλά προσθήκες που στόχο έχουν να τονίσουν κάποιες πτυχές. Δεν αλλάζουν όμως την γενική δομή του προγράμματος που προτείνει η Κομισιόν. Θα ήθελα να τονίσω ήδη τώρα ότι οι προτάσεις μου βασίζονται στην έρευνα για την υγεία, αλλά ε, ε, σχετίζονται και με άλλα θέματα που ενδιαφέρουν την ένδυ, ε, έστω και κάπως λιγότερα. Θα υποβάλω τροπολογίες ο ίδιος για τα θέματα που δεν είχα το χρόνο να εξετάσω αναλυτικά και ευχαρίστω θα εξετάσω προτάσεις των σχεδόν εισηγητών ή άλλων μελών της Επιτροπής μας. Όσον αφορά την, ε, τις έρευνες για την υγεία, ο στόχος είναι να ε, προωθηθεί η υγεία και η ευημερία όλων καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωής τους και είναι πολύ σημαντική η μετακίνηση από την θεραπεία στην πρόληψη και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την έρευνα ώστε να καταλάβουμε καλύτερα ε, τους παράγοντες της υγείας και τις ασθένειες που θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε καλύτερα προληπτικά μέσα συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων εμβολίων και ε, επίσης καλύτερες θεραπείες. Το, ε, επικροτώ το ότι η Κομισιόν τονίζει το θέμα των χρονίων ασθενειών που αυτή τη στιγμή επιβαρύνουν σημαντικά τα συστήματα υγείας μας. Ε, τα προβλήματα θα επιδεινωθούν στο μέλλον λόγω της γύρανσης ε, του πληθυσμού και γι' αυτό έχουμε την προστιθέμενη αξία της πρόληψης. Η Κομισιόν έχει συμπεριλάβει ε, παραδείγματα χρονίων ασθενειών, ο καρκίνος, οι ασθένειες της κυκλοφορίας κλπ. Ε, αντί να προσθέσω νέες ασθένειες ε, θα ήθελα να ε, διευκρινίσω ότι πρόκειται απλά για παραδείγματα τα οποία δεν προδικάζουν τις προτεραιότητες χρηματοδότησης της Κομισιόν στα προγράμματα. Αλλιώς θα καταλήξουμε σε έναν πολύ μακρύ κατάλογο ο οποίος ούτως ή άλλως δεν θα είναι εξαντλητικός, γι' αυτό νομίζω ότι είναι καλύτερο να διατηρήσουμε κάποιο βαθμό ευελιξίας. Μια πτυχή που πρέπει να τονιστεί περισσότερο κατά τη γνώμη μου είναι το τομέας των σπανίων ασθενειών και η ανάπτυξη των ορφανών φαρμάκων. Παρά την εσπανιότητά τους, οι ασθένειες αυτές ε, ε, ε, πλήττουν περίπου 30 εκατομμύρια Ευρωπαίους που δεν έχουν πρόσβαση σε θεραπεία επειδή σε κάποιες περιοχές δεν υπάρχουν, σε κάποιους τομείς δεν υπάρχουν θεραπείες. Ακριβώς εδώ θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιφέρει προσθέμενη αξία ενθαρρύνοντας την καλύτερη διάδοση των πληροφοριών και της γνώσης στον τομέα Αυτόν Θέλουμε ε, να ενθαρρύνουμε τα ε, προσωπικά φάρμακα τα οποία να είναι ε, προσαρμοσμένα στον γενετικό τύπο και τον τύπο ασθένειας του ασθενή του ασθενού. Έτσι μπορούμε να αποφύγουμε να ξοδεύουμε ένα σωρό χρήματα σε μη αποτελεσματικές θεραπείες. Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε τις ασθένειες που σχετίζονται με τη φτώχεια και θα πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την διεθνή συνεργασία στον τομέα αυτών. Επίση, πρότεινα στο σχέδιο γνωμοδότησης ε, σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος Ορίζοντα 2020 ε, να έχουμε ξεχωριστή προτεραιότητα για την περιβαλλοντική υγεία εντό του τομέα του περιβάλλοντο. Άσχετα από τον τομέα για τον οποίο μιλάμε, είναι σημαντικό να υπάρχει σχέση ανάμεσα στην επιστήμη και τις ε, κλινικές έρευνες ώστε να βεβαιωθούμε να μεταφέρονται τα αποτελέσματα, να μεταφράζονται τα αποτελέσματα σε καινοτόμα προϊόντα προ όφελο του συνόλου τη κοινωνία. Ε, γι' αυτό πιστεύω ότι το πρόγραμμα Horizon 2020 θα πρέπει να ε, στηρίζει την ε, διασυνοριακή έρευνα. Και επίσης πολλές χρόνιες ασθένειες έχουν παρόμοιους μηχανισμούς και η διασταύρωση πληροφοριών ανάμεσα στους διάφορους τομείς της ιατρικής μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με κάποιες ε, παρατηρήσεις για τα βλαστοκύτταρα, τα οποία εδώ και πολύ καιρό είναι επίμαχο κομμάτι της ε, πολιτικής ε, έρευνας και καινοτομίας. Καταλαβαίνω τα προβλήματα βιοηθικής και ότι οι εθνικές νομοθεσίες στο θέμα αυτό διαφέρουν. Ωστόσο, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις στο θέμα αυτό. Οι θεραπείες βλαστοκυτάρων έχουν ε, σημαντικά πλεονεκτήματα για τους ε, ασθενείς, ιδιαίτερα στην ε, αναγεννητική ιατρική ή ως θεραπεία για ασθένειες που απειλούν τη ζωή του ασθενούς. γι' αυτό σημαντικό είναι να στείλουμε θετικό μήνυμα τουλάχιστον όσον αφορά τα ενήλικα βλαστοκύτταρα ή τα εναλλακτικά εμβριονικά βλαστοκύτταρα, ακόμα και αν ε, θα πρέπει να αποδειχθεί η σχέση τους με τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα. Αλλά ε, θα μπορούσαμε να στηρίξουμε ε, τέτοιες πτυχές. Επίσης, ε, προτείνω αλλαγή στον τίτλο για να διασφαλίσουμε την κάλυψη των θεμάτων που σχετίζονται με τη διατροφή. Επίσης, μας ενδιαφέρει η έρευνα για τη βελτίωση της διατροφής και όσον αφορά το θέμα της ε, ενέργειας, ε, οι τροπολογίες ε, που προτείνω για τα δύο σχέδια γνωμοδοτήσεων στόχο έχουν να έχουμε πιο αποτελεσματικά και ανανεώσιμα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού και ε, και επίσης ε, προτείνω η αποδοτικότητα να αποτελέσει ε, μια πρόκληση ή έναν στόχο τον οποίο θα πρέπει να επιδιώξουμε σε όλο το πρόγραμμα Horizon 2020 όσον αφορά κάποια θέματα υλοποίησης. Σημαντικό είναι να έχουμε, σημαντικούς, να έχουμε σωστούς ε, σταθερούς δείχτες ε, για να αξιολογήσουμε την υλοποίηση του 2020 και να εξετάσουμε σε τι βαθμό η χρηματοδότηση ε, ανταποκρίνεται στους στόχους. Έχω υποβάλει κάποιες προτάσεις ε, σχετικά με τον ε, αριθμό θέσεων αποσχόλησης που δημιουργούνται, τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση και την συμβολή των μέτρων στην ανάπτυξη του ΑΕΠ. Επίσης έχω προτείνει κάποιες άλλες ε, τροπολογίες και μπορεί να υποβάλω ακόμα κάποιες. Ε, πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη για στρατηγικό συντονισμό ανάμεσα στις ε, έρευνες που χρηματοδοτούνται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να αποφευθούν οι επικαλύψεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Θα πρέπει τα προγράμματα έρευνα να επιφέρουν προσθέμενη αξία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συμπληρώνουν αυτά που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Τέλο, θα ήθελα να αναφερθώ στον προπολογισμό, που είναι ένα από τα, σημαντικότερα θέματα. Ε, όπω βλέπετε, δεν έχω υποβάλει τροπολογία σχετικά με τα νούμερα που προτείνει η Κομισιόν, πέρα από το 12% για τι έρευνε στον τομέα τη υγεία, ε, όπω άλλωστε ίσχυε και στο πρόγραμμα πλαίσιο 7, και μία δεύτερη τροπολογία που ζητάει περισσότερη στήριξη για τις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, η λύση που επέλεξα ε, έχει ε, επιλεγεί και από την αρμόδια της επιτροπή την Ήτρε και στόχο έχει να διασφαλίσει τη, σωστή χρηματοδότηση για κάποιους τομείς σε περίπτωση που αλλάξει ε, η πρόταση κατά τη συζήτηση του, των πολιτών, του δημοσιονομικού πλαισίου στο Συμβούλιο. Θα πρέπει να θα πρέπει να τα προσέξουμε τα θέματα αυτά αν θέλουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα και χωρίς να μπω αναλυτικά στον προϋπολογισμό θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ε, της έρευνας ε, και της καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πλήρη παρουσίαση της γνωμοδότησής σας. Τώρα έχουν το λόγο οι σκιώδεις εισηγητές. Θα σας παρακαλούσα να περιοριστείτε σε τρία λεπτά, διότι έχουμε ακόμα το θέμα live στην ημεροσία διάταξη και θα ήθελα να έχουμε αρκετό χρόνο για τη συζήτηση. Ε, Κουτιέρες Κορτίνες, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε παρέμβει μάλλον ε, έχουν μιλήσει κάποιοι σε προηγούμενα θέματα για 15 λεπτά και τώρα μας λέτε τρία. Τέλος πάντων. Εγώ εργάζομαι και στην Επιτροπή Ήτρε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρασπίσουμε όχι μόνο το περιβάλλον και την υγεία, αλλά και κάποιες αρχές, κάποιες γενικές αρχές ε, για την οργάνωση του προγράμματος ε, πλαισίου, ορίζον 2020. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε και τα δύο, και το περιβάλλον και την υγεία. Ένα παράδειγμα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ορισμοί για να μπορούν τα διαθροτικά ταμεία να χρηματοδοτούν την καινοτομία. Διότι τελικά η πράσινη οικονομία σημαίνει μεταβίβαση γνώσεων ε, και τεχνογνωσίας. Ευρωπαϊκή βιομηχανία δηλαδή. Πρέπει να δημιουργήσουμε στο πρόγραμμα πλαίσιο αλλά και στο σύστημα χρηματοδότησης ε, να προβλέψουμε πόρους για να μπορούμε να εργαστούμε και προς την κατεύθυνση του περιβάλλοντος και προς την κατεύθυνση της υγείας και θα πρέπει και οι περιφέρειες να δημιουργούν στρατηγικά σχέδια ε, που θα προωθούν την καινοτομία. Θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε υποδομές. Ορισμός ε, δεν υπάρχει για το τι εστί υποδομές. Δεν μιλάμε μόνο για υποδομές. Μιλάμε και για δίκτυα ασθενών, μπορεί να είναι και κάποια δίκτυα επικοινωνίας, ομάδες εργασίας για την πρόθεση της έρευνας. Είναι ιδέες που θα πρέπει να οριστούν, να οριστούν ξεκάθαρα σε όλα τα προγράμματα, για να μπορούν έπειτα να χρηματοδοτηθούν από τα διαδροτικά ταμεία. Εγώ θα πρόσθετα και το περιβάλλον. Επίσης και τις πράξεις δημόσιο δικού τομέα. Ο Ορίζον 2020 έχει ως εμβληματική πρωτοβουλία την, ε, ακριβώς της ΔΙΤ, την συνεργασία δημόσιο Δυτικού Μπορούν να γίνονται κλινικές, δομικές, ε, κλινικές δοκιμές από δημόσια νοσοκομεία με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, πολλές άλλες πρωτοβουλίες συνεργασίας δημόσιο τομέα. Όλα αυτά απαιτούν να έχουν υπόψη μας ότι θα πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό, να δώσουμε τη δυνατότητα να συμβεί. Και έχουμε και το συστημικό χαρακτήρα δεν μιλάω μόνο για, το διε, για τη διεπιστημονικότητα. Θα πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ κάποιων ε, εγκάρσιων ε, έργων και σχεδίων. Εγώ νομίζω επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μία έλλειψη. Επικεντρωνόμαστε μόνο στην αλλαγή του κλίματος. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για την εφαρμογή τεχνολογιών, για τη διαχείριση ε, των υδάτων, τον έλεγχο του υδροφορίζοντα και τέτοια θέματα. Και ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα που δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα είναι η επιστήμη και το πώς μπορεί να ε, επηρεάσει. Ας πούμε, η νευροεπιστήμη πρέπει να εφαρμοστεί στην παιδεία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η νευροεπιστήμη για την υγεία. Άρα, σχέση επιστημών και ε, εκπαίδευσης. δεν θα πρέπει στα παιδιά, παραδείγματο χάρη, να του ε, μαθαίνουμε πράγματα μόνο του παρελθόντο. Θα μπορούσαμε να τους διδάσκουμε ακόμη και τη γενετική γιατί αυτό βοηθάει και την λήψη αποφάσεων έπειτα από το πολιτικό σύστημα. Σε ό,τι αφορά την υγεία, δύο πράγματα και ολοκληρώνω. Πρέπει να επιμείνουμε στη διάγνωση, στη στήριξη για τη διάγνωση που είναι ουσιαστικά θέμα πρόληψης και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Πρέπει να στηρίξουμε τις προηγμένες ε, θεραπείες και την εξατομικευμένη ατρική. Ε, ο κάθε πολίτης, ε, ο κάθε ασθενής ε, θα πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται το μέλλον του. Και είναι μια ευθύνη που έχουν οι ασθενείς και αυτό θα πρέπει τις προηγμένες θεραπείες στην κυταρική και γενετική διάγνωση να τα προωθήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ που τηρήσατε τα τρία λεπτά. Ο Βιτόριο Πρόντιν, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, ή τον εισηγητή μάλλον, για την εισαγωγή και την εμβάθυνση στο θέμα. Οι προτινόμενες πρόκλησεις που περιέχονται στο νέο πρόγραμμα πλαίσιο για ανάπτυξη και έρευνα θέλουν να αυξήσουν την επιστημονική γνώση, να ενδυναμώσουν τη διάδοση των κέντρων αριστείας, να προωθήσουν τη βιομηχανική πρώτη θέση, να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις για να βρουν απαντήσεις στις μελλοντικέ προκλήσεις και στις ανάγκες της κοινωνίας για να εξασφαλίζεται η υγεία, ε, η ευημερία και η ασφάλεια των ατόμων και του περιβάλλοντος. Αφήνοντας κατά μέρος πτυχές γενικές που αφορούν τον προπολογισμό και διατάξεις ο καθορισμός των οποίων χρειάζεται πολύ λεπτομερή συνομιλία, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι πέρα από την εστίαση επιθεμάτων σημαντικών όπως η υγεία και η ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον δεν δέχεται επαρκή προσοχή. Η δράση για την αλλαγή του κλίματος και έχει έλλειψη, η έλλειψη πόρων και πρώτων υλών ε, έχει υποστηριχθεί λίγο έναντι των αναγκών και η καθαρή ενέργεια δεν τονίζεται ως ολοκληρωμένε μεταφορές. Όσον αφορά τη διάδοση των κέντρων αριστείας πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το όφελος να έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έρευνας ε, θα μπορούσε να προωθήσει προθυμένη έρευνα και αριστεία σε όλα τα κράτη-μέλη. Ιδιαίτερα δίνοντας προσοχή στο να μην τροφοδοτεί τις διαφορές μεταξύ ήδη κέντρων που είναι υποστηριγμένα από τα άλλα. Ε, θα πρέπει ε, να διατίθενται ανθρώπινοι πόροι και πόροι γενικά εκεί που χρειάζεται και να μην επιτρέπεται στις ίδιες προσωπικότητες να δέχονται νέα χρήματα και ήδη τα κέντρα αριστείας και τα πανεπιστήμια που υποστηρίζονται ή να επιστρέψουμε στα, κέντρα, ε, στα ίδια τα κέντρα αρχικά και να κολλάνε ιδέες. Λοιπόν, ε, η υποτροφία Μαρή Κιουρί είναι βασικός ε, ε, πόρος για την πρώτη ενέργεια και τη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου για την έρευνα. Όσον αφορά τις εργασίες αυτής της Επιτροπής, θα υποβάλω τροπολογίες που θα αφορούν την ανάγκη για μια έρευνα πιο εστιασμένη επί του περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα επί του εδάφους, διαχείρισης του εδάφους και έλεγχο των βιοτεχνολογιών, το διάστημα, ασφάλεια ε, τα γονιδιώματα και πιο γενικά την ε, προσωπική υγεία και τα προσωπικά φάρμακα. Θα, δεν προσέχουμε ένα θεμελιώδες στοιχείο. Τη διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Θεωρώ ότι δεν είναι προτεραιότητα και στη χώρα μου που ήδη έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και από σεισμούς για την καινοτομία έρευνα σαν εργαλείο ανταγωνιστικότητας. Αν θέλουμε το κοινό καλό, η έρευνα δεν θα πρέπει να οδηγεί μόνο σε εμπορικά ωφέλη, αλλά να οδηγεί σε πρόοδο κοινωνίας. Μία έρευνα που θέλει μόνο άδειε ευρεσιτεχνία και μετά δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματα αυτά σε εθνές επίπεδο, τροφοδοτεί μόνο τον κύκλο παραγωγής κατανάλωσης αποβλήτων ένας αυτοσκοπός που οδήγησε και στην παρούσα κρίση. Δεν είναι μόνο οικονομική κρίση και κρίση πόρων, αλλά και αξιών. Από την άλλη πλευρά, η ερεύνα για να διευκολύνει τη ζωή των ηλικιωμένων θα πρέπει να νικήσει ασθένειες όπως η Alzheimer και να μην και θα πρέπει τα ωφέλη τελικά να μπορούν να χρησιμοποιούνται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω έναν ε, επισκέπτη μας, ε, τον ε, Υπουργό Περιβάλλοντος της Κύπρου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαστε εδώ σήμερα μαζί μας και που μπορείτε να συμμετέχετε στην συνεδρίασή μας. Σας καλωσορίζω θερμά. Συνεχίζουμε. Η συνάδελφο Τζι Λέβεν, τρία λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ αναλυτική του εισαγωγή. Είναι πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά μπορούμε να συνδυάσουμε την έρευνα και την καινοτομία. Και αυτό πράγματι διανοίγει νέους ορίζοντες που θα μα επιτρέψουν να συμβάλλουμε στην ε, ανάπτυξη μια βιώσιμης και ανταγωνιστικής οικονομίας. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθεί η χρηματοδότηση σε αντικείμενα που είναι τη δική μα αρμοδιότητα, όπω ανέφεραν οι συναδελφοί, αλλαγή του κλίματο, ανώσιμε πηγέ ενέργεια, βιοποικιλότητα, υγειονομική περίθαλψη, ασφάλεια τροφίμων. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα κονδύλια αυτά θα πρέπει να συμβάλλουν στο στόχο της μείωσης ε, των, των εκπομπών διοξιδίου άνθρακα. Θα πρέπει να κάνουμε έρευνα για πιο μικρές αλυσίδες ε, τροφίμου και το καθεξής. Κάποια πρακτικά σχέδια και έργα που μπορούν όμως να κάνουν τη διαφορά. Και είναι και έργα που μπορούν να, να... στα οποία μπορούν να συμμετέχουν και μικρές επιχειρήσεις. Είναι ζωτική σημασία να είναι πιο προσβάσιμα τα κονδύλια αυτά σε μικρές εταιρείες Απαιτείται απλούστευση. Ο στόχος του 5% συμμετοχή περιλαμβάνεται στην νομοδότηση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι αγρότες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το στόχο. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που έχει ήδη αναφερθεί είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ευθυγράμμιση μεταξύ του ορίζοντα 2020 και των διαθροτικών ταμείων. Διότι με το συνδυασμό, τον αποτελεσματικό συνδυασμό αυτών των δύο μπορούμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα τη έρευνα και καινοτομία και των σχετικών βιομηχανιών. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία και τι διακρατικέ δράσει. Χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι στην νομοδότηση περιλαμβάνεται η αναπαραγωγική υγεία και το θέμα της ε, γονιμότητας. Ο αντίκτυπος ε, ε, του θέματος της υπογονιμότητας στην υγεία και στην καλή και στην ευεξία νομίζω ότι υποτιμάται κάποιες φορές. Εμεί είμαστε κατά το να χρησιμοποιούνται οι πόροι του ορίζοντα 2020 για τη χρηματοδότηση του ΙΤΕΡ, Νομίζουμε ότι μπορεί καλύτερα να αξιοποιηθεί η χρηματοδότηση για έργα ε, που μπορούν να έχουν απτά πραγματικά αποτελέσματα στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ώρα 2020 που θα βοηθήσουν να έχουμε μια οικονομία με αποτελεσματική χρήση των πόρων και χαμηλές εκπομπές του άνθρακα. Σας ευχαριστώ. Η Άννα Ρόσπαχ εκ μέρους της Γιούλη Κέρλινγκ. Καλά τα λέω. Καλά τα λέτε κύριε Πρόεδρε. Η σκιώδη συζητήτρια δεν μπορεί να είναι εδώ. Θα έρθει αργότερα. Οπότε στη θέση της θα κάνω εγώ μια σύντομη δήλωση η οποία αφορά και αυτή αλλά και την επόμενη έκθεση. Κύριε Γκέρλινγκ, γενικά είναι ικανοποιημένη με την πρόταση της Επιτροπής, διότι πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Απλά υπάρχουν θέματα που χρήζουν περαιτέρω εξέταση, Παραδείγματο χάρη, Πώ θα βρεθεί σωστή ισορροπία ε, για τη διαχείριση κινδύνου και την ε, επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων. πώ θα έχουν οι ΜΜΕ τη δυνατότητα να συμμετέχουν, να συμβάλλουν. Πάντω ε, και οι διεκθέσει πηγαίνουν προ σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη κάποια πράγματα ώστε η Ευρώπη να είναι στην πρώτη γραμμή της έρευνας και της καινοτομίας. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το ζήτημα είναι ουσιώδες. Η Επιτροπή μας, κατά την άποψή μου, πρέπει να δώσει έμφαση στην υγεία. Διότι σε αυτή την περίοδο πολύ σοβαρή κρίση που βιώνουμε, όταν πρέπει να γίνουν οικονομίε και περικοπές στον προπολογισμό, πολλές φορές δυστυχώς ο τομέας της υγείας είναι αυτός που πλήττεται. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε απόλυτα λέγοντας ότι η υγεία είναι προτεραιότητα για εμά, ε, στο πλαίσιο αυτού του πραγματοσπλαισίου. Και όχι μόνο για την ευεξία, ε, αλλά και ω πηγή ανάπτυξη. Αυτό άλλωστε λέγεται και στο πρόγραμμα που θα ψηφίσουμε το απόγευμα για την υγεία. Η έρευνα και η καινοτομία είναι ένα κλειδί της οικονομία. και πρέπει να το προβάλλουμε. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επίσης το λέμε πολλές φορές, υπάρχουν δυσκολίες. Πρέπει να πλουστευτούν οι διαδικασίες. Η ιατρική καινοτομία, επίσης πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόληψη Μίλησε για εμβόλια ο εισηγητή, αλλά έχουμε και την έρευνα για νέα αντιβιωτικά. Διότι εδώ έχουμε αντιμετωπίσει ένα πραγματικό πρόβλημα, μια πραγματική δυσκολία και πρέπει να επιμείνουμε στο θέμα, την ανάγκη δηλαδή για την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας και των νέων με ιατρικών τεχνολογιών. Συμφωνώ ότι δεν πρέπει να έχουμε ένα πολύ μακρύ κατάλογο. Μίλησε για σπάνιες ασθένειες ο εισηγητής φυσικά και θα τον υποστηρίξω Επίσης είναι σημαντικό να κάνουμε πάντο δυνατόν ώστε τα ερευνητικά εργαστήρια να παραμείνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Δυστυχώς ε, λόγω της κρίσης ίσως ε, μπουν στον πειρασμό να μετεγκατασταθούν σε άλλες χώρες. Θα πρέπει να θαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να καινοτομούν γιατί κάποιες φορές υπάρχει αδράνεια. Ξέρουμε ότι η καινοτομία στην αρχή κοστίζει αλλά στη συνέχεια μπορούν να εξοικονομηθούν με την καινοτομία πολλοί πόροι και ιατρική, ε, τα ιατρικά μηχανήματα είναι ένας πολύ ελπιδοφόρος τομέας για την καινοτομία. Και ολοκληρώνοντας υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ τόνωσης της έρευνας και της έκβασης, δηλαδή καινοτομία και πρόσβαση στην καινοτομία. Πρέπει να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα. Ωραίστε Ρώση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Πιστεύω ότι χρειάζονται περισσότεροι πόροι για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και πιο γενικά για να μπορούμε να ηγηθούμε βιομηχανικά και για την υγεία. Για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι πολύ λίγα η έρευνα. Μπορεί να δώσει πάρα πολύ μεγάλα αποτελέσματα σίγουρα και θα πρέπει να υποστηριχθεί με ιδιαίτερη προσοχή ε, όσον αφορά την πρόληψη σε αυτό το στοιχείο. Όπω το θέμα τη τεχνικής των γονιδιωμάτων ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα που έχουν οι πολίτες. Μπορούμε να έχουμε με πρόβλεψη πολύ έγκαιρη και να οδηγηθούμε σε καλύτερες συνθήκες ζωής για τα άτομα. Έχω τροπολογίες που θέλω να μειώσουν το κόστος της δίκης και διαχείρισης ώστε να βρούμε και άλλους πόρους χωρίς να αλλάξουμε τον προϋπολογισμό της νομικές επιχειρήσης και για την υγεία χωρίς να παρεύουμε επί του συνολικού αριθμού, αλλά αυξάνοντα και μετατίθεντε πόρους. Όσον αφορά τα βλαστοκύτταρα. Πολύ προσεκτικά το προσέξετε το θέμα ο Συγητή, ε, γιατί υπάρχουν και ηθικά προβλήματα όσον αφορά τα εμβριακά βλαστοκύτταρα. Θα πρέπει ε, να τα ανάκτηση των ομφαλίων λόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω αδυναμίας ε, μόνο το 1% των ομφαλίων λόρων ε, συλλέγεται με το θα μπορούσαμε να λύσουμε τα προβλήματα των ε, βλαστοκυτάρων, των βιακών χρησιμοποιώνταν τον ομφάλιο λόρο. Νομίζω ότι άλλα θέματα σαφέστατα αναφέρθηκαν από τον εισηγητή και νομίζω ότι είναι από τα σημαντικότερα νομοθήματα για τις μελλοντικέ εξελίξεις ε, στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση και την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή που σωστά εστιάζει στις χρόνιες ασθένειες. Πρέπει και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για τις ασθένειες αυτές. Επίσης, στην ε, στο πρόγραμμα, στην γνωμοδότηση, βρίσκω ότι ε, λείπουν έρευνες σχετικά με τις ε, ουσίες στο περιβάλλον μας που ε, επηρεάζουν τις ορμόνες και που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την υγεία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Oui, merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ έτσι να πω κάποια πράγματα για αυτή την πρόταση της ε, Κομισιόν. Ιδίω τα θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας. Φυσικά και πρέπει να προσανατολιστούμε προς μια πιο πράσινη οικονομία, αλλά αυτό τι σημαίνει εμείς ως πράσινοι δεν θέλουμε και μας είμαστε και αντίθετοι αυτό το πρόγραμμα ορίζων να μπορεί να χρηματοδοτεί προγράμματα όπως το ITER ή το Γκαλιλαίο. Η άποψη της ε, Επιτροπής και η πρόταση, κανονισμού βασίζονται πολύ στην τεχνολογία, ε, νομίζω, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα. Είναι η συμπεριφορά, η βελτίωση της κοινωνίας. Χαίρομαι λοιπόν που κατά κάποιο τρόπο υπάρχει ένα τμήμα για τις κοινωνικές προκλήσεις. Ασφάλεια τροφίμων. Γι' αυτό το σκέλος έχω να πω το εξής. Αναφέρεται ότι η παραγωγή ανθράκων θα πέσει σημαντικά τα επόμενα 40 χρόνια. Αυτό τι σημαίνει για τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων. Είναι πρόβλημα. Άρα πρέπει να προωθήσουμε μια πιο βιώσιμη και λιγότερη μικρότερη εξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες οικονομία. Φυσικά και θα πρέπει το αποτύπωμα άνθρακα να το μειώσουμε και την κατανάλωση να τη μειώσουμε βέβαια και έχουμε αυτή την πρόταση για μείον 20% μέχρι το 2020 και έχουμε και τα αέρια θερμοκηπίου. Λέμε ότι πρέπει να μειωθούν κατά 80% το 2050. Μήπως θα έπρεπε να ξεκινήσουμε ήδη από το 2035. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Ρίχαρτ Σίμπερ. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση του η γνωμοδότησή του συναδέλφου Μπουσό, ιδιαίτερα όσον αφορά τα, τις για τα βλαστοκύτταρα και την χρηματοδότηση. Αυτό ανταποκρίνεται ε, στις δικές μας πολιτικές ιδέες, ε, διότι θέλουμε τα κράτη-μέλη να έχουν ε, την δυνατότητα να θέσουν τις δικές τους ηθικές αρχές. Χρειαζόμαστε την έρευνα στην ε, κοινότητα για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το βιωτικό μας επίπεδο αυτή τη στιγμή. Ε, πραγματοποιείται η διάσκεψη Ρίο συν 20 και ε, τα θέματα αυτά είναι κεντρικά για το μέλλον όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και όλου του κόσμου. Θα ήθελα να εστιάσω στο θέμα του νερού και ε, την εταιρική σχέση ε, καινοτομία ε, που προβλέπει η Κομισιόν, ε, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκω τα απαραίτητα κίνητρα στην έκθεση. Η τεχνολογία του νερού μπορεί να συμβάλλει πολύ σημαντικά. Θα είναι ένα από τα κεντρικά θέματα, διότι οι πόροι εξαντλούνται και το πόσιμο νερό είναι κεντρικής σημασίας, όπως επίσης ε, και η ε, επεξεργασία των, ε, των υγρών αποβλήτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μέρκης. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που επέστησαν την προσοχή μας σε πολύ σημαντικά σημεία. Αυτό που με φοβίζει είναι μην έχουμε μια πολύ οριζόντια προσέγγιση ως προς αυτά τα θέματα. Θα έχουμε τελικά δηλαδή μια τέρμον κατάσταση, ένα κατάλογο θεμάτων θα πρέπει να ε, εξετάζουμε χωρίς να συσχετίζουμε αυτά τα θέματα μεταξύ τους. Νομίζω ότι κατά την άποψή μου υπάρχουν τρεις προκλήσεις κυρίως για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Αλλά αυτό που απαιτείται είναι να υπάρχουν γέφυρες, να υπάρχουν διασυνδέσεις, η υγεία. Παραδείγματος χάρη συνδέεται με το νερό. Ε, αν μιλάμε για το νερό, μιλάμε και για, τα, για τους ρήπους, ε, για τα διάφορα φωσφορούχα άλατα κτλ. Άρα πρέπει να έχουμε μια ε, προσέγγιση ολιστική και όχι σαλαμοποιημένη και στεγανοποιημένη. Πρέπει να βρούμε δηλαδή τους συσχετισμούς. Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η σχέση έρευνας και καινοτομίας δεν είναι αυτόματη. Η βασική έρευνα δεν καταλήγει απαραίτητο σε καινοτομία και είμαστε στην αναζήτηση, στην προσπάθεια αναζήτηση λύσεων. Γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε στι ευρωπαϊκές κοινωνίες μεγάλε προκλήσει. Αυτό όμω προσπαθούμε κυρίω να δημιουργήσουμε είναι νέε θέσει εργασία να επανεκκινήσει η οικονομία. Και αν θέλουμε να πετύχουμε, θα πρέπει να τονίσουμε το ρόλο των ΜΜΕ. Και με αυτό θα ολοκληρώσω. Εφιστώ την προσοχή σας όμως ακριβώς σε αυτό το σημείο. Πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις των καιρών μας. Άρα να βασιστούμε σε επιχειρήσεις μικρομεσαίες και στην έρευνα που έχει ως αντικείμενο της επιχειρήσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στον ορίζοντα 2020, στο πρόγραμμα Horizon 2020, πρέπει να σκεφτούμε βασικά το πώς μπορούμε να έχουμε αρκετά χαμηλά κατόφλια για τις συμμετέχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές που συνδέονται με τα ερευνητικά κέντρα του τομέα της υγείας. Να μην λαμβάνουμε μόνο υπόψη τα μεγάλα κονσόρτσια αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερον, θα περίμενα να εστιαστούμε περισσότερο στα τρόφιμα. Όχι μόνο την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά στα υγιεινά τρόφιμα, διότι η κατανάλωση τροφίμων σχετίζεται άμεσα με την υγεία και με τις χρόνιες ασθένειες. Τρίτον, θα συμπεριελάμβανα στις τροπολογίες μου περισσότερη εξέλιξη στον τομέα του εξοπλισμού και των εργαλείων και των δικτών για θεραπεία και αποκατάσταση ε, στο σπίτι και τα φάρμακα που χορηγούνται τακτικά. Διότι έχουμε ουρές σε όλα τα ιδρύματα της περίθαλψης στην υγεία και γι' αυτό πρέπει να έχουμε εξοπλισμό που είναι φιλικός προς τον χρήστη και έτσι να λύσουμε πολλά προβλήματα που να αντιμετωπίζονται στο σπίτι και να εφαρμόζονται και θεραπεία κατοίκων. Χρησιμοποιούμε υπολογιστέ σήμερα, χρησιμοποιούμε εργαλεία υψηλή τεχνολογίας. Καταλαβαίνουμε ότι χρειαζόμαστε κάποιες ε, οικιακές συσκευές υψηλή τεχνολογίας και θα έπρεπε, συνεπώς, να έχουμε περισσότερα από αυτά τα εργαλεία και από αυτού του είδου τον εξοπλισμό στο σπίτι για θεραπεία κάποιων ασθενειών. Όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιαστούμε επί των χρονίων ασθενειών, όπως είναι ο καρκίνος ε, και το Alzheimer και άλλες τέτοιες ασθένειες. Θα πρέπει επίσης να ασχοληθούμε και το θέμα της αντίστασης στα μικρόβια. Θα ήθελα να λάβετε λοιπόν υπόψη τις τροπολογίες που σας έχω υποβάλει. Ευχαριστώ πολύ Κρίστα Κλάς και μετά ο Πέτερ Λίζε. Δύο λεπτά καθένας. Ευχαριστώ πολύ. Σπάνια έχω δει να εργαζόμαστε τόσο σκόπιμα όσο σήμερα το πρωί. Όλοι έχουμε τον στόχο ε, κατά νου, αλλά μιλάμε για την έρευνα και θα ήθελα ε, να αναφέρω και την άλλη πτυχή, την ε, βασική έρευνα. Σημαντικό είναι η έρευνα ναι, ναι, ναι, η Ευρώπη να χρηματοδοτεί και την ε, βασική έρευνα. Η Ευρώπη μπορεί να το κάνει. Βλέπουμε όμως ότι τα πανεπιστήμια και τα ε, ερευνητικά ιδρύματα αγωνίζονται για την χρηματοδότησή τους και γι' αυτό οργανώνουν ε, προγράμματα ερευνητικά, αλλά να μην ε, κατακαιρματίσουμε τελείως ε, τον τομέα αυτόν. Η βασική έρευνα μπορεί να μας ε, φέρει νέα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσω υπέρ και της καλής χρηματοδότησης για τη βασική έρευνα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πέτερ Λίζε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον συντάκτη της γνωμοδότησης. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή η βάση αυτή για να επικεντρωθούμε στο θέμα της ε, έρευνας ε, στην υγεία. Ε, θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα την παρηγορητική γιατρική, τις σπάνιες ασθένειες και μαζί με την διατροφή. Μας ενδιαφέρει και το θέμα της υγείας των παιδιών. Ίσως θα πρέπει όμως να το θέσουμε πιο ευρέως το θέμα αυτό. Θα πρέπει να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την υγεία των παιδιών ε, και θα σας παρακαλούσα να συμπεριλάβετε και το θέμα των ε, προώρα ε, γεννημένων παιδιών. Όσον αφορά τον τομέα της βιοτεχνολογίας, η Κομισιόν ασχολείται και με το θέμα της της απομονωμένης διάγνωσης αλλά εγώ ως γιατρός ξέρω ότι η διάγνωση δεν με βοηθάει αν δεν έχω και ανάλογη θεραπεία Θέλουμε λοιπόν να στηρίξουμε την διάγνωση αν υπάρχει και θεραπεία. Βέβαια, μπορεί, δεν είναι πάντα δυνατόν αυτά να γίνονται ταυτόχρονα, αλλά θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Η τελευταία μου παρατήρηση έχει να κάνει με το θέμα της έρευνας στα βλαστοκύτταρα. Πιστεύω ότι είναι καλή θέση του εισηγητή. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτήν. Κάποιοι θα προχωρούσαν πιο πέρα, άλλοι θα τη θεωρούσαν υπερβολική, αλλά ε, μας ενδιαφέρει το θέμα των ε, αρμοδιοτήτων. Ε, ε, μας είπαν ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στις αρμοδιότητες της ΕΝΒΙ. Όταν μιλάμε για θέματα ηθικά, αυτά επίπτουν στις αρμοδιότητες της ε, Νομικής Επιτροπής. Ε, αλλά να το πω ως εξής. Δεν συζητάμε την ηθική πτυχή. Ο ε, η συγητής θέλει να τονίσουμε τις ε, δυνατότητες που προκύπτουν από την έρευνα στα βλαστοκύτταρα χωρίς ε, να ασχοληθούμε με τα ηθικά θέματα. Ε, θα υποβάλω σχετική πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος να δώσω το λόγο στην Κομισιόν και μετά στον εισηγητή. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι, διότι αμέσως μετά έχουμε το live και χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, καλωσορίζω όλα αυτά τα σχόλια που εκφράσατε και θα ήθελα να ξεκινήσω συμφωνώντας ότι δεν μας αρέσει ο σχηματισμός καταλόγων οι κατάλογοι έχουν αφαιρεθεί από τις συζητήσεις για την έρευνα στο Συμβούλιο. Έχει συμφωνηθεί να αφαιρεθεί ο κατάλογος, η λίστα, οπότε θα μπορέσει να υπάρξει πολεοτεμιακή προσέγγιση. Κάτι που απαιτείται για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της υγείας των πολιτών. Αντί να εξετάζουμε κάθε συγκεκριμένο πίνακα, κάθε ασθένεια ξεχωριστά, βλέπουμε ολιστικά τον ασθενή. Πρόληψη, πρόθεση, έγκαιρη διάγνωση, έγκαιρη θεραπεία. Θεραπεία λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά μας μελήματα. Όσον αφορά τα βλαστοκύτταρα, αναφέρθηκα σήμερα να τονίσουμε ότι η έρευνα για τα βλαστοκύτταρα είναι πολύ καινοτόμος τομέας έρευνας δείχνει να έχει μεγάλο δυναμικό και για τους ασθενείς και για τους ερευνητές και τους πανεπιστημιακούς και η θέση μας για τα πλαστοκύτταρα στο Horizon 2020 είναι να παραμείνει το status quo που ήταν ισορροπημένο, αποτελεσματικό, να συνεχίσουμε δηλαδή με τις ίδιες πρακτικές όπως με το οικονομικό πλαίσιο υπαριθμών 7 και το 6 δεν θα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, την έρευνα για τη δημιουργία στο ε, βλαστοκυτάρων, αλλά την έρευνα για τα βλαστοκύτταρα στις χώρες εκείνες, τα κάτι μέλη που δεν απαγορεύεται ρητά αυτή η έρευνα για τα βλαστοκύτταρα. Τώρα, οι αναφορές εναλλακτικά από τα εμβριακά βλαστοκύτταρα δεν είναι απαραίτητο, διότι στα κείμενα που υπάρχουν δεν αποκλείεται η χρήση τους και ίσως αν το αναφέρουμε ρητά ίσως να υπονομεύσουμε ανώτερα είδη. Αν είχαμε κατονομάσει τον, τα κύτταρα από τον ομφάλιο λόρο πριν ανακαλυφθούν άλλα ενήλικα στο κύτταρα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν θα είχαμε εμποδίσει αυτή την ανακάλυψη. παρόμοια διευκρινίσουμε τι χρηματοδοτείται και τι δεν χρηματοδοτείται ρητά, απλώς επαναλαμβάνουμε τα σαφώς δηλωθέντα. Δεν χρειάζεται αυτή η επικάλυψη. Για άλλες συγκεκριμένες ασθένειες και τεχνολογίες κρατήσαμε ευρείες αναφορές για να έχουμε προσέγγιση και εκ των κάτω προς τα άνω για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς ερευνητές και όλο τον κύκλο της καινοτομίας μέχρι τα νέα προϊόντα που θα αφορούν τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών. Για ίδιους λόγους δεν θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένα σημεία που αφορούν την ανανεώσιμη, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν χρειάζεται για να μπούμε σε συστήματα εναλλακτικά ενέργειας και βιώσιμα. Εδώ η σύλληψη και αποθήκευση του άνθρακα, η απόδοση, η ενεργειακή απόδοση κλπ. έτσι θα εξαιρούνται. Τόσο αφορά τι προτινόμενε αλλαγέ του τίτλου για την πρόκληση παριθμών 2 και να συμπεριλάβουν την ασφάλεια των τροφίμων, θα θέλαμε να πούμε ότι αυτό περιτεύει, διότι η ασφάλεια των τροφίμων συμπεριλαμβάνει ασφαλή ε, εφοδιασμό στην ασφάλεια των τροφίμων, τα ασφαλή τρόφιμα συμπεριλαμβάνονται. Όσον αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον, θεωρούμε ότι είναι εκτό πεδίο εφαρμογή, διότι εδώ αναφερόμαστε μόνο στη διαχείριση των θαλασσίων πόρων και όχι την ευρύτερη έννοια του γενικότερου θαλασσίου περιβάλλοντος. Τέλος, για τις ασθένειες που σχετίζονται με τη φτώχεια. Συμφωνούμε, ε, είμαστε υπέρ επεξεργασίας του θέματος, Φερρυπίν, η συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για τις κλινικές δοκιμές εστιάζεται, θα εστιαστεί πάνω σε αυτό το τομέα στο μέλλον. Ευχαριστώ την Κομισιόν. Πολύ σύντομα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά το πολύ χρειάζομαι να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση και σίγουρα θα συνεχιστεί. Καλωσορίζω την αναφορά στη διαχείριση των υδάτων που έκανε η κυρία Γκουτιέδες Κορτίνας, ο κ. Κάρας και η κυρία Μέρκης. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί ευπρόσδεκτες σχετικές τροπολογίες. Συμφωνώ με την κυρία Εύανς ότι θα πρέπει να τονίσουμε ε, τους πιο προσβάσιμους πόρους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η οικονομία με χαμηλές εκπομπές του άνθρακα πρέπει να είναι προτεραιότητα στις εργασίες μας. Προς τον κύριο Λίζε, ναι. Τα ηθικά θέματα δεν τα κάλυψα. Είμαι ε, αναπληρωματικό μέλος στη Νομική Επιτροπή και συμμετείχα στη συζήτηση. Ήθελα να τονίσω τις εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να υποστηριχθούν παρόλο που εξακολουθούν αυτά είναι τα θέματα για τη βασική έρευνα. Κυρία Κλάς, συμφωνώ ότι θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά σε αυτό διότι είναι σημαντικότατο για το μέλλον των ερευνών μας. Διεξάγεται μια συζήτηση για τα τρόφιμα, ότι χρειάζεται να εστιαστούμε περισσότερο στα τρόφιμα. Η κυρία Κούκοβετς το ανέφερε. Εγώ είμαι πολύ ανοιχτό, μπορώ να υποστηρίξω σχετικές τροπολογίες. δεν είχα περιθώριο και χώρο να καλύψω όλα τα θέματα, αλλά τα περισσότερα θέματα που συζητήθηκαν είναι πρόσδεκτα. Ευχαριστώ κυρία Γκροστέτ. Ε, έπρεπε, έβαλα την υγεία προτεραιότητα για την έκθεσή μου, είναι στο μέσο το ξέρω καλύτερα και συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις πρωτοβουλίες στον τομέα τη Υγεία και συμφωνώ απόλυτα και με τον κύριο Κοσένκο η ασφάλεια των τροφίμων θα πρέπει να καλύπτεται καλύτερα στην έκθεση ε, και στο πλαίσιο της καινοτομίας που συζητούμε. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρόντι και τον κύριο Ρώση. Για τον κύριο Πρόντι συμφωνώ με την πολιτισμική κληρονομιά, την πολιτιστική κληρονομιά. Επιτροπή Πολιτισμού θα ασχοληθεί με το θέμα και θα το στηρίξουμε όταν θα διεξαχθεί η τελική συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω θα παρουσιάσετε το χρονοδιάγραμμα και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την εκτίμηση που εξέφρασαν και ευχαριστώ την κυρία Λοξάνδρα Τάγκρακτη, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα λάβω υπόψη όλες τις προτάσεις της, τις αναφορές που έκανε και θα επιφέρουμε κάποιες αλλαγές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι αύριο. Στις 10 ε, Ιουλίου θα ξανασυζητήσουμε το θέμα εδώ στην Επιτροπή μας και στις 19 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια προβλέπεται για τον Νοέμβριο του 2012. Ε, αρμόδια επί της είναι η Επιτροπή Ήτρε και θα ήθελα να συμβολεύσω όλους τους συναδέλφους εάν θέλετε να ληφθούν υπόψη οι τροπολογίες σας υπάρχει η δυνατότητα να τις υποβάλλετε και στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. Υπάρχει και αυτή τη δυνατότητα. Παρακαλώ να το θεωρήσετε αυτό ως καλοπροαίρετη συμβουλή. Ε, ναι, ευχαριστώ. Θα λάβουμε υπόψη μας σε αυτήν την καλοπροαίρετη συμβουλή. Ε, αλλά εάν θέλουμε να συζητήσουμε εδώ με σοβαρό τρόπο, θα πρέπει να έχουμε και τη δική μας γνωμοδότηση θα παρακαλούσα μήπως μπορούμε να έχουμε μία ή δύο μέρες περισσότερες ε, τώρα ίσως ε, με τη ε, συζήτηση να έχουν προκύψει νέες ιδέες θα ήθελα να έχω διμερείς επαφές. μήπως μπορεί να παραταθεί η προθεσμία κατά μία-δύο μέρες, διότι από ό,τι γνωρίζω η Ήτρε θα ψηφίσει ε, αργότερα την, ε, την ε, σχετική έκθεση. Είναι κάτι που συνδέεται με τις δημοσιονομικές προοπτικές. Λίγο περισσότερο χρόνο μπορείτε να μας δώσετε. Ε, σας καταλαβαίνω. Και εμένα μου αρέσει να έχουμε χρόνο και να εργαζόμαστε σοβαρά πάνω στα θέματα, αλλά πληροφορίες που έχουμε λάβει μας λένε ότι δεν μπορούμε να αναβάλουμε την προθεσμία, αλλά θα το κοιτάξουμε. Με ενημερώνουν ότι αν παραλείψουμε την ανταλλαγή απόψεων τότε μπορούμε να ε, παρατείνουμε την προθεσμία. Τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να ψηφίσουμε. Εκτός εάν ε, συμφωνήσουμε να μην είναι απαραίτητα διαθέσιμες τροπολογίες, τότε το θέμα συνδέεται με την μετάφραση. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα. Ε, μία μέρα παράταση θα σημαίνει ότι θα λάβουμε τις ε, μεταφράσεις το Σεπτέμβριο. Ελπίζω ότι αν ε, ε, δώσουμε την Παρασκευή τις ε, τροπολογίες θα έχουμε μετάφραση τον Σεπτέμβριο, έτσι. Όχι, το θέμα είναι η συζήτηση στις 10 Ιουλίου. Σήμερα έχουμε 20 Ιουνίου. Εάν θέλουμε όλοι οι συνάδελφοι να έχουν τις τροπολογίες στη γλώσσα τους, θα πρέπει δυστυχώς να θέσουμε αύριο την προθεσμία όπως με ενημερώνει η γραμματεία. Δεν μπορώ να αφισβητήσω αυτό που μου λέει η γραμματεία. Εάν θέλουμε λοιπόν να μπορούμε να εργαστούμε εδώ με όλες τις γλώσσες θα πρέπει να τηρήσουμε την προθεσμία. Εάν δεν το θέλουμε αυτό, μπορεί να το αποφασίσει αυτό η Επιτροπή μας. Εάν δεν ε, τα θέλουμε όλα αυτά, τότε είναι δυνατόν να παρατείνουμε την προθεσμία για ε, τις τροπολογίες και να μην έχουμε στις 10 Ιουλίου όλες τις γλώσσες. Αυτές είναι οι δύο δυνατότητες. Πέτερ Λίζε. Ε, ναι, νομίζω ότι κατάλαβα τώρα. Ε, όταν ψηφίσουμε θα είναι απαραίτητο να έχουμε τις τροπολογίες σε όλες τις γλώσσες. Αλλά συζήτηση τον Ιούλιο ε, για ε, όλες τις τροπολογίες θα έχει νόημα ακόμα και αν δεν έχουμε τη μετάφραση σε όλες τις γλώσσες. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν μία-δύο μέρες προθεσμία ώστε τον Ιούλιο να μπορέσουμε να συζητήσουμε και τον Σεπτέμβριο να έχουν όλοι οι βουλευτές όλες τις τροπολογίες σε όλες τις γλώσσες. Gut, wir, der Vorschlag wäre Freitagmittag, dann haben wir... Προτείνεται προθεσμία Παρασκευή μεσημέρι για τις τροπολογίες με κίνδυνο για τη συζήτηση στις 10 Ιουνίου, ε, Ιουλίου να μην έχουμε τις ε, τροπολογίες σε όλες τις γλώσσες. Ε, Συμφωνία Επιτροπή. Βλέπω ιδιαίτερα τον συνάδελφο Λίζε να γνέφει καταφατικά. Λοιπόν, προθεσμία Παρασκευή μεσημέρι για υποβολή των τροπολογιών. Στις 10 Ιουλίου θα συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Ίσως να μην έχουμε τις τροπολογίες σε όλες τις γλώσσες και στις 19 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε και από ό,τι φαίνεται ε, τον Νοέμβριο συζήτηση και ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή, λέει ο Πρόεδρος, μάλλον στην Ολομέλεια εννοεί. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή. Περνάμε τώρα στο live. Το πρόγραμμα για το κλίμα και το περιβάλλον. Είναι ακριβό το πρόγραμμα αυτό. Και θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, Γιούτα Χάουκ, παραλίγο να πω στην ε, Υπουργό Οικονομικών μας. Ε, ναι, ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, το LIFE είναι μέρος της νομοθεσίας ε, των ε, πολιετών προγραμμάτων ε, που εμπίπτουν στο, πλαίσιο των νέων, στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και που μπορούν να βελτιωθούν. Στο παρελθόν το LIFE έχει αποδείξει την αξία του, οι εμπειρίες μας είναι καλές, είναι αποτελεσματικό το πρόγραμμα αυτό. Πολύ σύντομα ήταν ε, μεγάλη επιτυχία για όλους τους συμμετέχοντες ε, και αυτό το καταλαβαίνουμε όχι μόνο εδώ στην, ε, στο Κοινοβούλιο, αλλά και από περιφερειακές, τοπικές, εθνικές διοικήσεις, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ερευνητικά ιδρύματα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλοι επενούν το LIFE. Γενική επιτυχία λοιπόν και κυρίως κυρίες και κύριοι, είναι το μόνο μας πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών μέτρων. Έχοντας λοιπόν αυτό κατά νου, καθώς και την πρόκληση να έχουμε ε, μια βιώσιμη ε, κοινωνία, λέμε ότι θα πρέπει το σύνολο του προϋπολογισμού και όχι ε, μόνο το μικρό κομμάτι που αφορά το life, ε, να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το σύνολο του προϋπολογισμού ώστε να, ώστε να πετύχουμε τους ε, στόχους ε, Ευρώπη 2020. Θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου τους περιβαλλοντικούς στόχους. Θέλουμε λοιπόν με όλο τον προϋπολογισμό, θέλουμε όλο τον προϋπολογισμό να χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Υπάρχει το θέμα του mainstreaming, της το, το να συμπεριλάβουμε την βαλλοντική πτυχή σε όλα τα προγράμματα, αυτή είναι η μαγική λέξη. Όσον αφορά την ε, νομοθεσία, θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερις πτυχές. Την γεωγραφική ισορροπία, την ε, εθνική κατανομή δηλαδή, το ε, ποσοστό συγχρηματοδότησης, την δυνατότητα αποζημίωσης για το κόστος και τα ολοκληρωμένα προγράμματα. Ε, όσον αφορά το πρώτο θέμα, λοιπόν, ε, την ε, γεωγραφική ισορροπία, ήδη τώρα μας λένε συνέχεια η επιλογή των προγραμμάτων στις περιφέρειες γίνεται με βάση την ποιότητά τους και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους. Παρότι αυτό σημαίνει κυρίως επειδή αυτό το πολύπλοκο σύστημα επειδή έχουμε αυτό το πολύπλοκο σύστημα ε, ενδεικτικής εθνικής κατανομής, ε, αλλά αν κοιτάξουμε το ποσοστό υλοποίηση στα διάφορα κράτη-μέλη, βλέπουμε ότι κάποια κράτη-μέλη ξεπερνάνε κατά πολύ ε, τις ενδεικτικές τιμές, ενώ άλλα ε, δεν ε, τις φτάνουν κατά πολύ ή παραλίγο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και με ε, την εθνική κατανομή δεν ε, αποφεύγουμε τις ανισορροπίες. Εάν θέλουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, ξεκινήσουμε διαφορετικά. Τα κράτη-μέλη που έχουν χαμηλό ποσοστό έργων να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν προγράμματα υψηλής ποιότητας ε, και αυτό μπορεί να γίνει με εργαστήρια, ε, με εκπαίδευση και με την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με καλά επιτυχημένα προγράμματα. Ε, αυτό νομίζω θα είναι πραγματική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, το ποστό χρηματοδότηση στο παρελθόν, είδαμε ότι κάποια κράτη-μέλη ε, δυσκολεύονται με το ποσοστό συγχρηματοδότησης του 50%. Είχαν ε, δυσκολίες να βρουν το δικό τους 50%. Δεν ε, μπορούσαν να φέρουν το κόστος αυτό και εμείς θέλουμε ίση μεταχείριση όλων των κρατών μελών. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο, διότι κάποια κράτη-μέλη έχουν οικονομικές δυνατότητες, μια χαρά τα καταφέρνουν με το ποσοστό 50%, ενώ άλλα όχι. Και Γι' αυτό πιστεύω ότι με υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης ε, στις ε, οικονομικά πιο ασθενείς ε, περιφέρειες να πετύχουμε ισορροπία. Εάν σε όλους δώσουμε το υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης, αυτό θα σημαίνει ότι θα χάσουμε μια σειρά καλών προγραμμάτων. Ε, εάν πρέπει να δώσουμε δηλαδή 25% παραπάνω από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τότε θα έχουμε λιγότερα προγράμματα. Ε, ε θα έχουμε το, το, το, το ίδιο ποσό χρηματοδότησης αλλά όχι τον ίδιο αριθμό προγραμμάτων. Γι' αυτό η πρότασή μου είναι να παραμείνουμε στο 50% χρηματοδότησης ε, και στις ε, οικονομικά ασθενέστερες περιφέρειες ε, έχουμε παραμέτρους από την ε, διαρθρωτική και περιφερειακή πολιτική. Σε αυτές να δώσουμε το άλλο ποσοστό συγχρηματοδότησης. Επίσης όσον αφορά την επιστροφή των ταπανών. Η θέση της Κομισιόν είναι ότι με την αύξηση του ποσοστού χρηματοδότηση, ε, να μην μπορούν να αφαιρεθούν ε, ε, οι δαπάνε για το μόνιμο προσωπικό και το ΦΠΑ. Ιδιαίτερα το δεύτερο σημείο είναι προφανές για μένα, διότι αν δούμε τον ταπεινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μας και εκεί μέσα το ταπεινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE Ε, και από εκεί το ΦΠΑ πηγαίνει στο Ταμείο των Περιφερειακών ε, Τοπικών Εθνικών Αρχών, ε, ότι με το ΦΠΑ αυτό χρηματοδοτούνται τα ταμεία αυτά. Αυτό το βρίσκω λάθος. Αλλά ποια είναι η λογική. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι τοπικές και εθνικές αρχές μας εξηγούν ότι α, όχι δεν γίνεται, αυτό θα είναι απόλυτη καταστροφή αν το καταργήσουμε. Θα αποτύχουμε και δεν θα μπορούμε να ε, πραγματοποιήσουμε προγράμματα live. Η πρότασή μου είναι, όσον αφορά το ΦΠΑ, να ε, τηρήσουμε τον ε, Γενικό Δημοσιονομικό Κανονισμό. Εκεί λέει οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και άλλοι ε, μη δημόσιοι φορείς Το κράτος μέλος όπου δεν επιστρέφεται ε, ο ΦΠΑ, ε, επιστρέφεται ο ΦΠΑ από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Ε, κατά την επιστροφή των, των ταπανών για το μόνιμο προσωπικό αυτή η επιστροφή πιστεύω ότι θα πρέπει να περιοριστεί στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Με κανέναν τρόπο δεν θα ήθελα πανεπιστήμια, πόλεις ε, ή περιφερειακές αρχές να χρηματοδοτούνται με τον τρόπο αυτόν. Ε, και φτάνω στο ε, τέταρτο μου θέμα, τα ολοκληρωμένα έργα. Όποτε περνάει ο πρόεδρος από το γραφείο μου φωνάζει από την πόρτα ολοκληρωμένα έργα. Τα ολοκληρωμένα έργα είναι ένα νέο μέσο. Αλλά η ιδέα είναι εξαιρετική κατά τη γνώμη μου. Αν πάρουμε την ε, ευρύτερη βάση, ε, κοιτάξουμε τι έχουμε. Έχουμε το νερό, το περιβάλλον, ε, το κλίμα. Υπάρχουν ταμεία με περισσότερους πόρους από το LIFE. Αν ε, αυτά τα ταμεία τα συμπεριλάβουμε ε, στο πρόγραμμα μας, ε, το Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης, το, το Ταμείο για την Ανάπτυξη της Πέθρου, το Ταμείο για την Αλληλεία, αυτά έχουν περισσότερα χρήματα από το πρόγραμμα LIFE μας. Ε, μιλάμε λοιπόν για συγκεκριμένα μέτρα mainstreaming, για τη συμπερίληψη της περιβαλλοντικής πτυχής στα προγράμματα αυτά. Εάν εισάγουμε αυτή την πτυχή του LIFE σε αυτά τα προγράμματα ε, για, τα οποία είναι αρμόδια επί της ουσίας σε τα άλλα ταμεία, θα μπορέσουμε ε, να τα συνδυάσουμε. Το αν και πώς θα λειτουργήσει αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Ε, άλλωστε δεν είναι και αυτό το καθήκον μας. Εμείς ε, θέλουμε να ξεκινήσουμε υποχρεωτικά. Ε, άλλωστε ο κόσμος ε, ανήκει στους τολμηρούς. Κλείνοντας ε, να πω ότι η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί κατά τη γνώμη μου πολύ καλή βάση υπό τη μορφή που έχει για τις συζητήσεις μας και τη λήψη αποφάσεων ε, αναμφισβήτητα, αλλά ε, στο κοινοβούλιο ισχύει αυτό που ισχύει και στην πραγματική ζωή, ότι το καλύτερο είναι εχθρό του καλού. Ε, εγώ προτείνω 60 τροποποιήσεις στο κείμενο της Κομισιόν και φαντάζομαι ότι και οι συνάδελφοι θα έχουν καμιά δυο ιδέες ακόμα σχετικά με το τι μπορούμε να αλλάξουμε στο κείμενο της Κομισιόν. Περιμένω εναγωνίως να ακούσω τις θέσεις σας. Ε, νομίζω ότι όλοι μπορέσατε να διαβάσετε την ε, πρότασή μου εκτός από τους γερμανόφωνους, ε, διότι το γερμανικό κείμενο δεν το έχουμε λάβει. υπάρχει όμως το κείμενο σε όλες τις άλλες γλώσσες. οι Γερμανοί θα το διαβάσουν μετά. Ευχαριστώ Γιούτα Χάουκ για την παρουσίαση της... Ε, παρουσίαση έκθεσής σου με τον μοναδικό σου τρόπο και ε, περνάμε τώρα στους σκιώδεις εισηγητές ε, και θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα ε, στο σκιώδη εισηγητή του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Βέβαια μας στηρούσε ενήμερους ε, ανα πάσα στιγμή κατά την εκπόνηση της έκθεσής της. Οπότε πρέπει να πω ότι αυτά που είπε στην εισαγωγή της με βρίσκουν σύμφωνοι. Είχα και ενημερωθεί βέβαια ότι είναι ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα που πρέπει να συνεχιστεί. Συμφωνώ με την εισηγήτρια που μιλά για το mainstreaming και την ε, σωστή χρήση των πόρων. Σε ό,τι αφορά τα ολοκληρωμένα έργα, integrated projects, και εγώ στην αρχή δυσκολεύτηκα να καταλάβω περί τίνος πρόκειται, όταν όμως είδα τα έγγραφα, άρχισα να καταλαβαίνω κάπως καλύτερα. Από ό,τι κατάλαβα, πρόκειται για έργα που έχουν προχωρήσει, έχουν ολοκληρωθεί, νεοτορισμός αυτός, καινοτομία, αλλά είναι χρήσιμα μόνο όταν δεν απορροφούν κονδύλια από άλλα έργα. Σίγουρα πρέπει να ορίζονται καλύτερα στην νομοθετική πράξη, όπως λέει η συγγήτρια. Δεύτερον, γραφειοκρατία. Έχω συζητήσει αυτό το θέμα με τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι θα ήθελαν η διαδικασία υποβολή των ε, υποψηφιωτήτων να είναι ταχύτερη και η διαδικασία λήψεως αποφάσεων να είναι απλούστερη, πιο γρήγορη και βέβαια και η υποβολή των αντισοπληρωμής και η καταβολή των πληρωμών να είναι ταχύτερη και απλούστερη διαδικασία. Τώρα, χρηματοδότηση Υποστηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεγαλύτερη χρηματοδότηση 70 και 80% σε ορισμένες περιπτώσεις. Νομίζω ότι είναι μια καλή πρόταση. Συγχρόνως όμω, αν λάβω υπόψη τι πληροφορίε που έχω λάβει, έχω υπόψη μου ότι είναι δύσκολο να βρεθεί χρηματοδότηση για έργα στον τομέα τη βιοπικιλότητα. Μήπω θα έπρεπε να χρηματοδοτήσουμε και αυτά τα έργα με 70%. Τώρα, γεωγραφική ισορροπία και κατανόμη των σε επίπεδο. Δεν συμφωνώ με την άποψη της Ήτρες ω προς αυτό το σημείο. Νομίζω ότι είναι καλό να υπάρχει αυτή η εθνική κατανομή όπως υπήρχε μέχρι τώρα. Και να μην περιορίζεται αυτό στο ολοκληρωμένο έργο όπως προτείνει η Κομισιόν. Υπάρχουν λόγοι και επιχειρήματα που συνηγορούν προ αυτήν την κατεύθυνση. Ήδη ίδια η Επιτροπή Ευρωπαϊκή στα πρώτα χρόνια της εφαρμογής του προγράμματος LIFE δεν περιμένει πολλά έργα. Το ένα τρίτον πρέπει να είναι μάλλον παραδοσιακά. Και ένα άλλο επιχείρημα που αναφέρει η συγκήτρια είναι ότι η εθνική κατανομή είναι ένα ενδεικτικό στόχο ε, για την άντληση κονδυλίων από τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ποιότητα του έργου διακυβεύεται. Η ποιότητα του έργου και η διάθεση εθνικών πόρων συμβαδίζει. Και είμαστε υπέρ του να παραμείνουν αυτοί οι πόροι. Eh, eh, σε ό,τι αφορά τώρα την έννοια της αλληλεγγύης, έχουμε κάποιες σκέψεις. Προτείνεται η έννοια αυτή να αντικαταστεί ε, σε, εθνικούς, ε, το, τα national allocations. Υπάρχουν διαφορετικοί ρυθμοί ανάπτυξη στα διάφορα κράτη-μέλη. Εδώ μιλάμε για ένα πρόγραμμα όπου η ποιότητα έχει στη σημασία. Έχουμε προγράμματα όπως το Horizon 2020, το COSME και άλλα. Και το πρόγραμμα απευθύνεται σε αναπτυγμένες και λιγότερο αναπτυγμένες ε, χώρες. Η προσέγγιση αυτή λοιπόν φαίνεται λίγο αμφισβητήσιμη. Η χρηματοδότηση των κρατών μελών στο πλαίσιο του LIFE πιστεύω ότι θα πρέπει να καθορίζεται σε συνάρτηση με το βαθμό ανάπτυξης αυτού του κράτους μέλους. Και κάτι άλλο που ανέφερε η συγγήτρια είναι ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη το κόστος μόνιμο προσωπικό ΦΠΑ. Νομίζω ότι είναι σωστό ότι πρέπει να προωθήσουμε την ισότιμη μεταχείριση. Γι' αυτό και συμφωνώ με την πρόταση για το ΦΠΑ. Σωστό είναι να στηρίξουμε και την απασχόληση, τη μόνιμη απασχόληση προσωπικού, να μην υπάρχει ανάγκη δηλαδή ανάθεσης υπηρεσιών σε υπεργολαβία και κάποια τεχνικά σχόλια. Πρόγραμμα εργασίας, από ό,τι προβλέπετε προς το παρόν, διετής θα είναι η διάρκεια. Μήπως θα έπρεπε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να επιμικρύνουμε την περίοδο για το πρόγραμμα εργασίας. Γιατί απαιτείται μεγαλύτερη χρηματοοικονομική σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τους παρόχους. Σε ό,τι αφορά τη μουσεία, φαίνεται ότι λείπει το έδαφος. Είναι σημαντικό όμως. Δεν υπάρχει αυτή η ιδέα εδώ και θα έπρεπε να περιλαμβάνεται. Επίσης πιστεύω ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να δίνει έμφαση στην υλοποίηση. Όλο, όλα τα προγράμματα, όλα τα έργα πρέπει να κατατείνουν ακριβώς αυτό, στην υλοποίηση προγράμματα στον τομέα της ε, πληροφόρησης, επικοινωνίας, ε, αύξησης της ευαισθητοποίησης, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, θα πρέπει να θεωρείτε ότι είναι υποστηρικτικά προ άλλα προγράμματα. Σα ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Πρέπει να προσέξουμε τον χρόνο, διότι έχουμε άλλο ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη, το οποίο πρέπει να προλάβουμε να συζητήσουμε. Ε, θέλουμε να ακούσουμε και την Κομισιόν. Ε, αν δεν έχετε αντίρρηση, προτείνω να περιοριστούμε στα 2,5 λεπτά ο καθένας και να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Chris Davis που εκπροσωπεί τον συνάδελφο και Παρακαλώ. Προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Συμφωνώ με την εισηγήτρια. Το live το αγαπάμε, είναι επιτυχημένο, θέλουμε να παραμείνει. Ε, πράγματι για να αυξηθεί ο προπολογισμό του αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να αφαιρεθούν πόρια από αλλού. Επίσης θέλουμε να υπάρχουν πιο πολλά ολοκληρωμένα έργα για να έχουμε την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας τιμής, προστασία τα κτλ. Είμαστε προετοιμασμένοι να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο απάψη πια εθνική κατανομή και να ανταγωνίζονται τα κράτη-μέλη για να αποδείξουν ότι τα προγράμματα που ε, προτείνουν το αξίζουν. Αξίζουν να πάρουν τη χρηματοδότηση. Πιστεύω ότι αν ξέρουν ότι υπάρχουν πόροι θα είναι πρόθυμα τα κράτη-μέλη να ε, υποβάλουν και σωστούς φακέλους και να υποβάλουν ποιοτικά προγράμματα για τη χρηματοδότηση. Ο συνάδελφος Κεμπράντη δεν ε, είναι πεπισμένος για το ότι πρέπει να αυξηθεί το σκέλος της χρηματοδότησης σε περιθωριακές περιοχές τομείς. Δεν είμαι εγώ προσωπικά βέβαια απόλυτα βέβαιος, ίσως να έχει δίκιο η συγγήτρια Καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες που θα εφαρμόζονται παντού. Και ότι πράγματι αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση σε κάποιες περιοχές ή χώρες μπορεί και να μην εκτελειωστούν καν ε, τα έργα. Και επειδή κάποιες οργανώσεις όπως η BirdLife Life ε, ασκούν κάποιες πιέσεις ώστε να διατηθούν πόροι ε, και για τα υπερπόντια εδάφη και διαμερίσματα της Ένωσης, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη βιοπικιλότητα, είναι μια ιδέα που με βρίσκει σύμφωνο, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα, αυτό είναι το πρόβλημα. Ο προπολογισμό είναι πολύ μικρός. Εγώ θα προτιμούσα ίσως να είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί ένα έργο εξαιρετικό, αν θέλετε. Να μην κλείσουμε εντελώς την πόρτα, αλλά εν γέννη δεν μπορώ να το στηρίξω διότι αν Απλώς, αν θέλετε τη μαρμελάδα σε ακόμα μεγαλύτερη φέτα, θα είναι ακόμα πιο λεπτή η στρώση. Ευχαριστώ. Έχουμε και μια ομάδα επισκεπτών από την Βιντσέντζα. Ο Σνάφος Μπελάτο έχει και προσκαλέσει την ομάδα επισκεπτών αυτή. Τους καλωσορίζουμε. Gut, es geht weiter. Als nächstes hat dann die Kollegin Προχωρούμε. Τζούλι Γκέρλινγκ, επόμενη ομιλήτρια, για δυόμιση λεπτά, παρακαλώ. Thank you and uh, may I add my congratulations to the report. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να προσθέσω τα συγχαρητήριά μου προς την εισηγήτρια. Ε, πραγματικά με πολύ μεγάλη χαρά εργάστηκα και εγώ για αυτήν την έκθεση. Δύο-τρία σημεία πολύ γρήγορα. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε εδώ να οριστικοποιήσουμε τα περί του προπολογισμού μέχρι ισότου ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει στο Κοινοβούλιο εν γέννη. Αλλά στηρίζω την άποψη τη εισηγήτρια και τη Κομισιόν ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο προπολογισμό του LIFE. Και είναι προτεραιότητα λόγω και των περιορισμών που υπάρχουν σε σχέση με την αλλαγή του κλίματος. Τώρα υπάρχει ένα κενό χρηματοδότηση, παραδείγματο χάρη για του τόπου ε, Natura 2000, ίσω θα μπορούσαμε το mainstream για την περιβαλλοντική χρηματοδότηση να το αξιοποιήσουμε σε άλλα προγράμματα πιο αποτελεσματικά και να βρούμε μια ικανοποιητική λύση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έξυπνη ε, η πρόταση για το ΦΠΑ. Έχουμε και το κόστος, ε, τη δυσκολία από το επιλέξιμο κόστος, το μόνιμο προσωπικό. Όλα αυτά θα τα στηρίξουμε πάντως εμείς. Στηρίζω επίσης ε, για μέτρα ε, δημιουργίας υποδομών, capacity building σε κράτη-μέλη που δεν έχουν υψηλά ποσοστά απορρόφησης. Στηρίζω την πρόταση, αλλά για την αντικατάσταση του συστήματος των ενδεικτικών εθνικών κατανομών δεν συμφωνώ να καταργηθεί αυτό το σύστημα. Προτιμώ να διορτηρηθεί, όπως είπε και η συνάδελφο Ρωμάνα Τζόρτ. Μήπως ο πανευρωπαϊκός ανταγωνισμός, αυτή η προοπτική αποθαρρύνει μικρές μικρομεσαίε επιχειρήσεις να καταθέσουν προτάσεις. Δεν νομίζω λοιπόν ότι έτσι θα αυξηθεί η ποιότητα, όπως λέει η συγγήτρια, ίσως έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Και απαντώντας στα σχόλια για τα ε, περπόντα εδάφη και διαμερίσματα Chris Davis. Εγώ συμφωνώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει επίπτωση στον προπολογισμό. Πάντα θα κρίνονται με βάση τα υπέρ και τα κατά τα έργα. Μην βάλουμε κάτι ακόμη στο μείγμα, γιατί ε, ενώ είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα χρηματοδοτηθεί κάποιο υπερπόντιο ε, έργο, καλό θα ήταν να υπάρχει, να αναφέρεται πάντως. Γκατιέρες Κουτίνες. Δύο λεπτά και τριάντα δεύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Η Γιούτα Χάουκ ε, πραγματικά αποτελεί εγγύηση, ε, ιδίως για αυτό το θέμα, γιατί έχει μια ευρωπαϊκή νοοτροπία η Γιούτα και αυτή η επανακρατικοποίηση του Life εμένα με ανησυχεί. Στην προηγούμενη εκδοχή του Life ήμουν σκιώδης εγώ και υπήρξε μπλοκάρισμα του Life, όλοι οι βουλευτές. Χρειάστηκε να περάσουν 8 ε, μήνες για να μπορέσουμε να περάσουμε τη χρηματοδότηση. Οι χώρες δε είχαν λάβει ήδη αποφάσεις τους εμείς συσχετίσαμε την ποιότητα με την Ευρώπη και προασπίζαμε την ποιότητα. Κάποια κράτη-μέλη όμως ενέκριναν έργα στα οποία επαναλαμβανόνταν τεχνολογίες που ήταν, ε, είχαν ανακαλυφθεί εδώ και χρόνια. Δεν ε, βρισκόταν κάτι καινούριο, μα το live σημαίνει καινοτομία. Άρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναλαμβάνουμε μελέτες, τεχνολογίες, προτάσεις. Αυτή είναι η ταυτότητα του live και οι χώρες που τα πήγαν καλά και ήταν ανταγωνιστικές τελικά κατάφεραν να κερδίσουν περισσότερους πόρους από αυτούς που θα λάμβαναν αν είχαν επανακρατικοποιήσει τα έργα, όπως η χώρα μας. Πήραμε 20 εκατομμύρια ευρώ και η κυβέρνησή μου με κατέκρινε γιατί εγώ την κατηγορούσα με τα προγράμματα που θα έπαιρνε 20 εκατομμύρια. Με τα προγράμματα όμως που κατέθεσε πήρε 36 τελικά εκατομμύρια. Κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι ένα σχήμα το οποίο υπάρχει μέσα στο σχέδιο και υπάρχει κατά της καρτικοποίησης. Η φύση δεν έχει σύνορα ούτε όρια. Ένα ποτάμι ε, δεν ανήκει στη χώρα από την οποία ε, περνάει, αλλά σε όλες τις χώρες από, την οποία, από τις οποίες περνάει. Μιλάμε για την ε, ρήπανση των θαλασσών, το, μιλάμε για τη μείωση εκπομπών κτλ. Αν θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε το οικοσύστημα και αν βασιστούμε στις γνώσεις που ξέρουμε και τις επιστημονικές γνώσεις, δεν μπορούμε να προωθούμε εθνικά έργα. Πρέπει να επιτρέπουμε να αναπτυχθούν διακρατικά έργα. Μελέτη των πτηνών. Όταν τα πτηνά μεταφέρονται, από, πηγαίνουν μάλλον από την ε, Σουηδία στην Αφρική, ούτε άδεια ζητάνε, ούτε βίζα. Θα διαβάσω πολύ προσεκτικά τις τροπολογίες βέβαια και προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι τροπολογίες που ενδεχομένως θα καταθέσω. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν θέλουμε σύνορα, ούτε ελέγχου στα σύνορα στον τομέα του περιβάλλοντος. Ε, θέλουμε ένα καλό πακέτο και καλή υλοποίηση των προγραμμάτων. Ε, μας αναφέρατε το παράδειγμα της Ισπανίας ε, που υλοποιεί πολύ καλά τα προγράμματα αυτά. Ε, τελευταία στον κατάλογό μου είναι η Λίντα Μακέβαν. Παρακαλώ. Um, Θα είμαι πολύ γρήγορη. Ευχαριστώ τη Γιούτα για την ευελιξία που έδειξε για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις μόνιμες συμβάσεις πολλοί πρέπει να επιβιώσουν έχοντας ε, συνεχάς επιμονήμων έργων κάποιους να ασχολούνται. Ευχαριστώ για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Απευθύνομαι εν μέρη προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω έναν, ε, ένα μέρο τη εκλογική μου περιφέρειας ε, που είναι μικρομεσαία επιχειρήση και ήθελε να είναι υποψήφιο το Life. Αλλά είδε ότι είναι μικρή εταιρεία μόνο μετά από ένα εξάμεινο πέντε πρώτη πληρωμή και μετά από 11 μήνε τους υπόλοιπου πληρωμές. Κανονικά όλε οι μικρομεσαίες επιχειρήσει θέλουμε να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα. Με το Life τι γίνεται. Διότι όπως λέει ο εκλογέας μου στην επιστολή του δεν μπορεί να περάσει έξι μήνες χωρίς να έχει κάποια πληρωμή, χωρίς καμία πληρωμή. Ευχαριστώ Λίντα. Να δώσω σύντομα το λόγο στην Κομισιόν. Ποιο θα ήθελε να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Κομισιόν. Euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω καταρχάς την εισηγήτρια, την κυρία Γιούτα Χάουγκ, για το σχέδιο εκθέσεώς της και για τις τροπολογίες που έχουν σαν στόχο να προταθούν βελτιώσεις επί του κειμένου και επί διαφόρων σημείων αυτού. Θα αναφερθώ σε κάποια στοιχεία. Κυρίως θα αναφερθώ σε αυτά που είπε η κυρία εισηγήτρια και οι βουλευτές. Ξεκινώ από την έννοια της γεωγραφικής ισορροπίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της, όπως υπογραμμίσατε, θέλησε να πετύχει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να συνεχιστεί το πρόγραμμα LIFE, που με μέτριο προϋπολογισμό που σε πεσημάνθη είχε τεράστια επιτυχία και υποστηρίχθηκε και από τα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή τη ήθελε να προσεγγίσει το πρόγραμμα LIFE, αυτό το μετριοπαθέ στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών και καταπολέμηση αλλαγή του κλίματος, αλλά ταυτόχρονα θα χρησιμοποιήσει καλύτερα το πρόγραμμα αυτό, ούτω ώστε να συμπεριλάβει περιβαλλοντικές πτυχές και καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών στι άλλε κοινοτικέ πολιτικέ και στα ολοκληρωμένα έργα θέλαμε να ευθυγραμμιστούν οι διάφορε πτυχέ με αυτά που υπόθηκαν πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα οι εθνικέ ε, κατανομέ για να γίνεται σεβαστή η γεωγραφική κατανομή στα κάτι μέλη των πόρων. Έχουμε 20 χρόνια εμπειρία όσον αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων και είδαμε όπω υπογραμμίστηκε από την κυρία Συγήτρια ότι η έννοια τη Εθνική διανομή έστω και ενδεικτική δεν επέτρεπε πάντα την επίτευξη των στόχων τη κατανομής αυτή. Όπω αναφέρθηκε κάποια κάτι μέλη είχαν μεγάλη επιτυχία και εφάρμοσαν πολλά προγράμματα και απορροφούν κοινοτικούς πόρους του LIFE, ενώ άλλες χώρες παρά τις προσπάθειες που έγιναν σε εθνικό επίπεδο δεν τα κατάφεραν να πετύχουν την ποσόστοση που τους ανήκε σύμφωνα με το σύστημα εθνικών κατανόμων και τα προγράμματα που ήταν ποιοτικά, έξοχης ποιότητας, ε, δεν εφαρμόστηκαν ε, λόγω της ε, κακής αυτής της εθνικής κατανομής. Γι' αυτό δεν προτιμήσαμε στην πρότασή μας αυτή την προσέγγιση και θέλαμε να έχουμε τα ποιοτικά κριτήρια. Όμως δεν θέλω να επισημάνω ότι η πρόταση της εισηγήτριας, δηλαδή να υποστηριχθούν περισσότερο τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για να εφαρμόσουν τα προγράμματα όσον αφορά την κοινοτική χρηματοδότηση, μια προσέγγιση για να αποφύγουμε το εθνικό σύστημα κατανομής, έστω και ενδεικτικό, να εφαρμόζεται που καμιά φορά ε, είναι μια μεταβλητή παραπάνω για τα προγράμματα και τα έργα. Κάτι άλλο που αναφέρθηκε είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της ήθελε καταρχάς να πλουστεύσει την κατάσταση, να πλουστεύσει ε, τις εκθέσεις, της χρηματοδότηση, να πλουστεύσει τον περιορισμό των δαπανών, κυρίως τον φόρο επί του ΦΠΑ και το κόστος του μονίμου προσωπικού, απλουστεύοντας δηλαδή να, να μην αυξάνοντας τη συγχρηματοδότηση για να μην επιβαρύνουμε ε, τους ετούντες. Στο πνεύμα της απλούστευσης κάναμε διευκολύνσεις και καλύτερη διαχείριση. Στην υποβληθήσα πρόταση να ξεχωριστά να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά οι μειονεκτούσες περιοχές, ε, μας δημιουργήθηκαν προβλήματα εφαρμογής. Πώς καθορίζονται οι λιγότερο ευνοϊκές περιοχές. Πέρα από τα προγράμματα που θα ασχολούνται με αυτές τις περιοχές, που θα διαχωρίζουν τις περιοχές ευνοϊκές από τις μη ε, ευνοϊκές, ε, πρέπει να δούμε και τι γίνεται με το πεδίο εφαρμογή του προπολογισμού όσον αφορά το LIFE. Ίσως χρειάζεται περαιτέρω προβληματισμός, αλλά ήδη διαβλέπουμε προβλήματα εφαρμογή και δυσκολίες και διερωτώμε πού θα γίνει αυτό. Δεν είναι μέσω συνοχή το LIFE που θα εφαρμοστεί αυτή, αυτό το προτιμησιακό καθεστώ για τι λιγότερο ευνοημένε περιοχέ. Όσον αφορά τα ολοκληρωμένα έργα, σημειώνω με θικανοποίησο την υποστήριξη τη σχεδόν ομόφωνη που διαπιστώθηκε για τα ολοκληρωμένα έργα που επισημοποιούν για πρώτη φάση του περιπολογισμού του LIFE την, το πτυχή μόχλευση των μικρών περιβαλλοντικών προγραμμάτων LIFE ε, με τα άλλα προγράμματα που χρηματοδοτούν πολύ περισσότερο. Άρα μπορούμε να έχουμε και εδώ φιλοδοξίες πολύ μεγαλύτερες όσον αφορά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου για το περιβάλλον που απαιτεί αυτό και μια προσπάθεια. Αναφέρθηκαν και θέματα των υπερπεριφερειακών περιοχών και τα εδάφη, τα υπερπόντια. Αυτά αναφέρονται και σε άλλες επιτροπές. Εκεί που συμμετείχαμε σε ανάλογες συζητήσεις δεν μπορώ παρά να επενθυμίσω το μικρό προπολογισμό που διατίθεται για το πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να καλύψουμε μεγάλη επικράτεια. Όλα εξαρτώνται από μελλοντικέ αποφάσεις, δημιουργείται και πρόβλημα διαχείρισης Έχουμε την εμπειρία του προγράμματος για τις τρίτες χώρες που συμπεριλαμβάνονταν στο προηγούμενο live, το live 3, και εκεί αντιμετωπίσαμε τεράστια προβλήματα εφαρμογής, κυρίως όσον αφορά την ανάκτηση των κοινοτικών πόρων και υπενθυμίζω το στόχο του προγράμματος που είναι να υποστηρίξουμε οικονομικά την εφαρμογή των πολιτικών. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ναι, ναι, τώρα τελειώνω, λέω. Ε, σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, Κάθε περιφέρεια που δεν εφάρμοζε το κοινοτικό δίκαιο όσον αφορά το περιβάλλον δεν μπορούσε να υποστηριχθεί με τον δεδειγμένο τρόπο. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει εναλλεκτικέ λύσει ενδεχόμενε όσον αφορά τους πόρους ε, ανάπτυξη. αν μπορούμε να βελτιώσουμε εν αυτή τη ενία την πρότασή μα. Ευχαριστώ. Ζήτω συγγνώμη που Έπρεπε να σας διακόψω τόσο απότομα, αλλά έχουμε και ένα άλλο θέμα στη μέση διάταξη. Ε, δεν απαντήσατε στην ερώτηση της Λίντα Μακέβαν ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 30 δευτερόλεπτα, αν μπορείτε. Ή μήπω ε, να το λύσετε διμερός και να δώσω πολύ σύντομα το λόγο στην ε, εισηγήτρια. Ε, τις, ε, όσον αφορά τις πληρωμές όταν ε, συμμετέχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι στον προϋπολογισμό μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ε, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, θα το κοιτάξω, αλλά αν έχουμε την προθεσμία των τριών μηνών, Εν πάση θα το κοιτάξω, θα δω πώ είναι το θέμα αυτό. Ευχαριστώ όλου του συναδέλφου που πήραν το λόγο. Πολύ σύντομα όσον αφορά ε, τα OTC. Και εγώ καταλαβαίνω ότι κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Όλοι όσοι αναφέρονται στο τομέα της ανάπτυξης και συμμετέχουν στο JPA ε, θα ε, πρέπει να φροντίσουν ε, ώστε να εκμεταλλευτούμε και το EDF για να προωθήσουμε προγράμματα βιοπικιλότητας. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση, Judy Gerling. Καταλαβαίνω, σε εποχές λιτότητας θα πρέπει παντού να κάνουμε οικονομία και γι' αυτό λέτε ότι δεν θα πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος. Αλλά δεν μιλάμε για πραγματική αύξηση. Η αύξηση αυτή δικαιολογείται απόλυτα από τα, τις νέες αρμοδιότητες του ΛΑΕΦ. Το κλίμα ε, και τα ολοκληρωμένα προγράμματα ουσιαστικά δεν πρόκειται ήδη κατά την πρόταση της Κομισιόν ε, για αύξηση. Αλλά να σας το πω εξής. Εγώ δεν έχω κλείσει το θέμα ε, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να μας δώσουν παραπάνω από όσα ζητάει η Κομισιόν. Εγώ σκέφτομαι ότι με λίγα δημόσια πίεση θα μπορέσουμε να πάρουμε λίγο περισσότερα ώστε ε, να μπορέσουμε με 10% να μπορέσουμε να στηρίξουμε όλες τις ε, περιοχές μας Natura 2000 και γι' αυτό δεν χρειαζόμαστε 3,2 δισεκατομμύρια, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 5,3 για μια 7 ετία. Και αν το υπολογίσετε αυτό δεν είναι πάρα πολλά. Τελεία. Ευχαριστώ πολύ, Γιούτα Χάουκ. Προθεσμία για την υποβολή των απολογιών 24 Ιουνίου στις 12. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, θα ψηφίσουμε 17-19 Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ για το θέμα αυτό στη ημερησία διάταξη και τώρα φτάνουμε στο θέμα 8 της ημερησίας διάταξης. Ε, έχει να κάνει, πρόκειται για μια ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 ε, του κανονισμού REACH. Ε, η απαγόρευση της χρήσης του μολύδου και των ενώσεών του σε κοσμήματα και εξαρτήματα για τα μαλλιά. Πρόεδρε, μπορούμε να επανέλθουμε μετά το γεύμα και να ψηφίσουμε κάτι. Τεράστια δουλειά έγινε για την προετοιμασία φακέλων, αποδείξεων λοιπά επιστημονικών. Τεράστια ποσά μπήκαν. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε το θέμα σε 3,5 λεπτά. Είναι απαράδεκτο. Δεν γίνονται αυτά. Ich möchte Richard Seber das Wort geben. Der hat nämlich... Να δώσω το λόγο στον Ρίχαρτ Ζήπερ. νομίζω ότι ο Κριστέιβε έχει δίκιο, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε σε 3,5 λεπτά. Δεν ε, ξέρω τι έγινε με την ημερησία διάταξη. Νομίζω στι 5 η ώρα έχουμε τον κύριο Ταγιάννη. Ε, δεν ξέρω αν η Γραμματεία πράγματι πιστεύει ότι από τις 3 έω τι 5 θα ψηφίζουμε επί δύο ώρε. Μήπω υπάρχει εκεί λίγο περιθώριο και να περιμένει ο Επίτροπος ε, ένα τέταρτο και να το συζητήσουμε αυτό το απόγευμα. Ε, να ξεκινήσουμε ακριβώ στι 3 προτείνω ώστε να έχουν όλες... Ε, να μπορούν να πάρουν σωστά το λόγο όλοι οι συνάδελφοι. Έχει δίκιο ο Χριστέβης. Ναι, καταλαβαίνω την ένσταση του Κρίς. Λίντα. Ναι, συμφωνώ. Θέλω να ακούσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσω το πώς θα ψηφίσουμε. Αν συζητήσουμε το θέμα στις 3, θέλω διάλειμμα πριν ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε, πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα αυτό το θέμα στην Επιτροπή. Δεν θέλω να έχω συζήτηση και μετά ψηφοφορία. Θέλω χρόνο να συμβουλευτώ με το συζητήσω με συναδέλφους που ψηφίσω. Πρόταση έχουμε το θέμα αυτό ως πρώτο στις ψηφοφορίες στις 3 η ώρα. Θα μπορούσαμε να έχουμε την ψηφοφορία στο τέλος και να δούμε τι θα γίνει με το χρόνο. Αυτή είναι η πρότασή μου, διότι έχει δίκιο. Η Λίντα Μακέβαν θέλει να ακούσει την ε, Επιτροπή και να έχει κάποιο διάλειμμα πριν την ψηφοφορία. Μπορείτε να δεχτείτε αυτή την πρόταση, ο Ρίχαρτ Τζέιμπερ. Παρακαλώ να έχουμε αρκετό χρόνο για τη συζήτηση, διότι στο θέμα αυτό είχαμε πάρα πολύ πίεση από τα λόμπι και θα πρέπει ε, να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Οι διαδικασίες ε, σχετικά με το θέμα αυτό ε, ήταν απίστευτες. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο που χρειαζόμαστε για να το συζητήσουμε αυτό. Προτείνω λοιπόν στι 3 ώρα να ξεκινήσετε τι ψηφοφορίε, τον υπόλοιπο χρόνο να τον ε, εκμεταλλευτούμε για τη συζήτηση. Να ακούσουμε την Κομισιόν, ε, διότι πρέπει να το συζητήσουμε τώρα, ε, να το ψηφίσουμε, διότι μας πιέζουν τα λόμπι. Πρόταση, να ακούσουμε τώρα την Κομισιόν, να δώσουμε τώρα το λόγο στην Κομισιόν για το θέμα αυτό. Φρανσουάζ Κορτέτ και πάντα με αυτέ τι αλλαγέ των προγραμμάτων τελευταία στιγμή. Ξέραμε ότι είχαμε διάφορα θέματα να επεξεργαστούμε το πρωί. Ίσως πρέπει να τα χειριστούμε διαφορετικά από την αρχή. Αυτό είναι το πρώτο. Διότι κάθε φορά το ίδιο πρόβλημα έχουμε σε κάθε επιτροπή. Δεύτερον, όταν λέμε ότι υπήρχαν πιέσει στον λόμπι, λυπούμε. Αυτό αφορά εταιρείε με παγκόσμιο φήμη στη Γαλλία και δεν είδα ούτε ένα λόμπι. Εξεπλάγιν με αυτό που λέει ο Αυστριακό συνάδελφο. Νομίζω ότι υπήρχαν ε, λόμπι σε κάποιους, ε, λόμπι από κάποιου βουλευτέ που έγινε. Να πρέπει να λέμε την αλήθεια καμιά φορά. Πρέπει να πω ότι πάνω σε αυτό θα πολεμήσουμε. Διότι παίρνει μια καμπή απαράδεκτη εδώ, μια τροπή απαράδεκτη. Απ' την άλλη πλευρά Υπάρχουν συμφορίες που πρέπει να ξεκινήσουν στις 3, πρέπει να γίνουν κανονικά. Εγώ ζήτησα μια χάρη, δεν ζητώ συχνά χάρες. Η έκθεσή μου να περάσει πάρα πολύ γρήγορα. Μου είπαν ε, δεύτερη νομίζω. Συμφωνούσε συνάδελφος, αλλά απουσιάζει την έσω αυτή τη στιγμή. Αλλά αρκετά πια με αυτή την ανοργανωσιά της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Υγείας. Κυρία Γκουτιέρεφ, ε, θα πω κάτι πολύ απλό. Αυτό ε, το έγγραφο το έχει προωθήσει ένα λόμπι. Οι ρυθμιστές τελικά παίρνουν ενδείξεις από τους ρυθμιζόμενους. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και είναι και πια και τόσο κατεπήγον. Θα χαθεί ο κόσμος εάν ε, δεν ε, ψηφίσουμε αμέσω. Αν δεν γίνουμε λιγότερο γραφειοκρατικοί και δεν συζητήσουμε αυτό το ζήτημα το σοβαρό, δεν πρέπει να υπάρχει το κριτήριο της δικαιοσύνης, της ενημέρωσης και της ισότητας. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ακαδημαϊκή, είμαι πανεπιστημιακή και αρνούμε να ψηφίσω κάτι χωρίς να το έχω συζητήσει. Και υπάρχει και ένα θέμα δεοντολογίας και ηθικής. Θέμα υπευθυνότητα. Δεν θα ψηφιστεί αυτή η έκθεση αν δεν τη συζητήσουμε wollen wir auch nicht heute. Wir werden sicherlich nicht sterben. Ε, όχι, δεν θέλουμε να πεθάνουμε σήμερα, είτε το συζητήσουμε είτε όχι, αλλά έχουμε το θέμα αυτό στη μερίσια διάταξη. Συζητήσαμε τον κανονισμό, ακούσαμε επικρίσεις. Πρέπει σήμερα να ψηφίσουμε. Προτείνω λοιπόν να αφήσουμε την ημερήσια διάταξη ως έχει, να το ψηφίσουμε πρώτο, προτού να ψηφίσουμε όμως να ακούσουμε την Κομισιόν και να μην υπάρξει συζήτηση. Μα πρέπει να γίνει συζήτηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, είτε θα το συζητήσουμε τώρα, χωρίς διαρμηνία... Εδώ και δέκα λεπτά συζητάμε τον την ημερήσια διάταξη και τον κανονισμό. Ξέρω από κάποιες ε, ε, ομάδες ότι δεν έχουν πάρει ακόμα θέση. Θέλουν πρώτα να ακούσουν την Κομισιόν. Οι εκπρόσωποι της Κομισιόν είναι παρόντες, είναι προετοιμασμένοι. Έχουμε το θέμα 8 στην ημερησία διάταξη. οι συνάδελφοι ε, έχουν ε, διατυπώσει αυτή την ένσταση, πρέπει να τη συζητήσουμε, πρέπει να επεξεργαστούμε. Είναι πολύ κανονική ε, διαδικασία αυτή. Ε, πάντα μια χαρά τα καταφέρουμε το χρόνο στην Επιτροπή μας. Αυτό που λέτε ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο δεν ισχύει και άλλωστε ο καθένας νομίζει ότι είναι ο πιο σημαντικός και θέλει να πει τη γνώμη του. Προτείνω χωρίς διερμηνία να το συζητήσουμε, αλλά η κυρία Σατουχάση έχει ένα διαδικαστικό. Ε, νομίζω ότι είναι απαράδεκτο. Ο μόνος που επιτρέπεται να μιλήσει είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπρόσωπο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον μία παρέμβαση για κάθε ομάδα. Να διεξαχθεί συζήτηση. Linda. Η Λίντα. Αν έχουμε χρόνο από διερμηνία να ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ψηφίσουμε στις τρεις, στις κανονικές εκθέσεις μετά συζήτηση για το θέμα που ακούσαμε να αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά δεκάλεπτο διάλειμμα και μετά ψηφίζουμε μπορούμε να αναβάλουμε για τις 5.30 να έρθει στις 5.30 ο κ. Σταγιάννη και συνεχίζουμε αργότερα τη συζήτηση. Να ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα έχουμε χρόνο να σκεφτούμε κατά τη του γεύματο, μετά συζητάμε το απόγευμα και μετά δεκάλεπτο διάλειμμα ψηφίζουμε. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό. Διότι θα πρέπει να συζητήσουμε, είναι σημαντικό θέμα και νομίζω ότι θα χρήσιμο να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα, όπω προτείνει ο Πρόεδρο. εάν δεν υπάρχει αντίρρηση, να ακούσουμε την Κομισιόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσουμε να πω ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθνικών Σώων εκπροσωπείται εδώ από τον κύριο Βανιού. Αν λοιπόν έχετε ε, στην υπηρεσία να απευθύνετε συγκεκριμένα ερωτήματα, κάντε το. Το πρώτο που θα θέλαμε να αναφέρουμε είναι μια υπενθύμηση. Ποιος είναι ο στόχος ε, του περιορισμού που συζητείτε. Θέλουμε να προστατεύσουμε την ανθρώπινη υγεία και συγκεκριμένα των νέων παιδιών από επικίνδυνες συνέπειες ε, των, ε, του μολύβδου σε διάφορα κοσμήματα. Ε, διότι σύμφωνα στοιχεία τα νέα παιδιά μπορούν να εκδίδονται ε, μέσω λόγω του τρόπου συμπεριφέρονται και με τα πράγματα βάζουν στο στόμα τους κινδυνεύουν τα παιδιά. Η πρότασή μας δεν καλύπτει μόνο τα αντικείμενα για τα νέα παιδιά, αλλά και αντικείμενα για τους ενήλικες. Το λέω αυτό διότι υπάρχει μια επίκριση που ακούγεται που λέει ότι ο περιορισμός μας αφορά δεν συγκρίνεται με τον ΙΠΑ. Συγκρίνεται με τον ΙΠΑ και μάλιστα είναι ευρύτερος, ευρύτερο το πεδίο που καλύπτουμε από τη ΣΥΣΥΠΑ. Η πρόταση περιορίζεται, απαγορεύει τη χρήση ε, μολύβδου στα κοσμήματα και τη διάθεση αυτού των αντικειμένων στην αγορά αν περιέχουν μόλυβδο σε μια συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,05% και έχει κάποιες εξαιρέσεις εσωτερικά ρολογιών, φυσικές πέτρες, δεν μπορεί να φάει το εσωτερικό ρολογιό ένα παιδιού, αντικείμενα μεταχειρισμένα όσο είναι πάνω από 50 ετών και εξαίρεση που συζητείτε το μολύβι που βρίσκεται μέσα σε κρυστάλλινα ποτήρια. Σε... Δεν μιλάμε για πολυελαίους, δεν μιλάμε για μαχαιροπίνα και διάφορα πράγματα στο τραπέζι. Τρεις επικρίσεις έχουν ακουστεί όσον αφορά την πρότασή μας, όσον αφορά το σχέδιο και τις εξαιρέσεις. Πρώτα απ' όλα ότι η κοινωνικονομική αξιολόγηση που έγινε από διάφορη επιτροπή, η επιτροπή πρότεινε κάποιες εξαιρέσεις ενώ δεν υπάρχει μελέτη για τον αντίκτυπο, για την υγεία. Άλλοι επίκριση ότι θα μπορούσε στα κρυστάλλινα ποτήρια χρησιμοποιηθεί εναλλακτική εκτός μολύβδου με τα ίδια οπτικά και φυσικά χαρακτηριστικά και τρίτη επίκριση αφορά το ότι η εξαίρεση που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ευρύτερη από τη σύσταση της κοινωνική Επιτροπής Αξιολόγησης και επεκτείνεται σε όλα τα κρυστάλλινα ποτήρια και όχι μόνο σε δύο από τα τέσσερα από τις τέσσερις κατηγορίες. Κάτι που θα πρέπει να αναφερθεί για τις εξαιρέσεις είναι ότι εδράζεται επί της απουσίας σημαντικού κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και βασίζεται και στην έλλειψη στοιχείων εναλλακτικών για το μόλιβδο. Ε, πρώτα απ' όλα ο κίνδυνος. Η απουσία σημαντικού κινδύνου ήδη αναγνωρίστηκε στο, αρχικό φάκελο που υπέβαλε ένα κάτω μέλος, η Γαλλία συγκεκριμένη περίπτωση, ε, δεν αμφισβητήθηκε από την, αξιολόγηση, από την Επιτροπή Αξιολογήσεως Κινδύνου, δεν αμφισβητήθηκε και όταν η Επιτροπή αυτή ασχολήθηκε με το θέμα, παραδέχτηκε το γεγονός ότι υπήρχε έλλειψη διαθεσίμων στοιχείων για σημαντικό κίνδυνο. Σημείωσε επίσης ότι το να βάλει κανείς τα κρυστάλλινα ποτήρια στο στόμα δεν σημαίνει ότι απελευθερώνεται μόλιβδος και άρα δεν υπήρχε σημαντικός κίνδυνος. Επ' αυτής της βάσης, εφόσον η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι επιφορτισμένη με την αξιολόγηση της αναλογικότητας, ε, μπορεί να κάνει κόστος ωφέλους, ανάλυση κόστος ωφέλους. Ε, το όφελος είναι μηδενικό, οδήποτε κόστος πάνω από το μηδέν θα ήταν κάτι δυσανάλογο. Αν υπάρχει έλλειψη λοιπόν αποδείξεων σημαντικών ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος, εν τη αυτή περίπτωση κανένα μέτρο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ενδεδειγμένο μέτρο. Η Κοινωνική Επιτροπή Αξιολόγησης δεν ξεπέρασε τα όρια της εντολής που δόθηκε, έκανε την ανάλυση κόσοφέλους που απαιτεί εντολή που δόθηκε για να αξιολογήσει την αλογικότητα. Εναλλακτικέ λύσεις. Λέει εναλλακτική λύση που ταιριάζει, αυτή που είναι εφικτή οικονομικά και τεχνικά. Εννοούμε, τεχνικά εφικτή. Η Επιτροπή είπε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, ότι υπάρχει ε, εναλλακτική που ταιριάζει στην αγορά. Λέει επίσης ότι οι εναλλακτικές ίσως να μην προσφέρουν την ίδια διάχυση του φωτός στο κρίσταλο όπως το μολύβι και ότι ίσως να μην προσφέρονται και όλα τα διαθέσιμα χρώματα για το κρίσταλο. Ας πούμε το χρώμα του ρουμπινιού. Η εναλλακτική, ποια άλλη ήταν, ε, ότι λιγμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας η ύπαρξη ενός τέτοιου δεν σημαίνει ότι μια διαδικασία είναι διαθέσιμη εκτός εργαστηρίου ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανική κλίμακα. Ένας κατασκευαστής ίσως είχε τη δυνατότητα να παράγει γυαλί παρόμοιας ποιότητας χωρίς μόλιβδο. Λέμε χωρίς μόλιβδο, διότι αν δεν έχει μόλιβδο δεν είναι κρίσταλο. Γι' αυτό λέμε γυαλί χωρίς μόλιβδο. Αλλά από ό,τι ξέρουμε σε άλλους εμπορευόμενους δεν είναι θεσιμή τεχνολογία. Πέραν αυτού δεν είχαμε πληροφορίες που να δόθηκαν κατά τις διαβουλεύσεις όσον αφορά τις φυσικές χημικές ιδιότητες των εναλλακτικών λύσεων, πώς μπορεί να γίνει η επεξεργασία, ποια είναι η σκληρότητά τους, ποια είναι η βιωσιμότητα των υλικών αυτών. Αυτές τις γνώσεις έχουμε τώρα. Προβλέπεται και ρήτρα αναθεώρησης διότι γνωρίζουμε ότι θα μπορούσε να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τα στοιχεία, τις τεχνολογίες για τις εναλλακτικέ. Γι' αυτό έχουμε ρήτρα αναθεώρηση πέντε χρόνια για να έχουμε χρόνο για πληροφορίες και για να επιτευχθεί τεχνολογική πρόοδος. Τρίτη επίκριση, όπως προανέφερα, αφορούσε την επέκταση εξαίρεσης της ΣΕΡΚ από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπόθηκε ότι για ηλεκτρονικό εξοπλισμό ε, είχαμε τέσσερα είδη κρυστάλλων που εξαιρέθηκαν και εμείς πήραμε όχι μόνο τους δύο της ΣΥΡΚ αλλά και άλλες δύο κατηγορίες βάλαμε. Να υπενθυμίσω έλλειψη σημαντικού κινδύνου για τις δύο κατηγορίες οι οποίες αρχικά αξιολογήθηκαν και αυτές οι δύο κατηγορίες είναι αυτές που περιέχουν τη μεγαλύτερη ποσότητα του μόλιβδου. Αν υπάρχει έλλειψη σημαντικού κινδύνου λοιπόν, όταν υπάρχει μεγάλη περιεκτικότητα σε μόλιβδο, εξορισμού, χαμηλότερη περιεκτικότητα ε, σημαίνει ακόμα χαμηλότερο κίνδυνο. Και επεκτείναμε αυτή την εξαίρεση για λόγους συνοχής σαφήνειας στην ομοθεσία έχοντας επίγνωση ότι δύο ε, νομοθετήματα διαφορετικά δεν έχουν τον ίδιο σκοπό αλλά είναι πολύ πιο πρακτικό η εμπορευόμενος να έχουμε εξαιρεσει που καλύπτουν τον ίδιο τομέα. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Αυτή η προσέγγιση έτυχε ομόφωνη υποστήριξη επιτροπή REACH, δηλαδή και από τα 27 κράτη-μέλη, εν κατακλείδη το σχέδιο πρότασης για τους κινδύνους και για παγόρευση για τα κρίσταλα με μόλιβδο λόγω ελήψεως αποδείξεων για κίνδυνο στην ανθρώπινη υγεία εν τη απουσία τεκμηριωμένων εναλλακτικών λύσεων διαθεσίμων στην αγορά και σε έναν τομέα για τον οποίο γνωρίζουμε ότι χαρακτηρίζεται από πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα δεν θεωρούμε ότι αυτή η προσέγγιση θα ήταν ανάλογη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Κομισιόν. Αυτά που μόλις μας εξηγήσατε ήδη έχουν υποβληθεί γραπτός στους συναδέλφους. Μπορούν λοιπόν να τα εξετάσουν. Να δώσω σύντομα το λόγο στην ε, υπηρεσία, στον Οργανισμό Χημικών, παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η απάντηση που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει τις βασικές στοιχείες. Η Επιτροπή Ανάλυσης παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία και δόθηκαν και γραπτός απαντήσεις. Εξετάστηκε η συνέπεια για την υγεία σε συνεργασία με την Επιτροπή Εξολογήσεως Κινδύνου. Και οι δύο επιστημονικές επιτροπές το εξέτασαν το θέμα. Εντελεχέστατα. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλοι οι συνάδελφοι θα ενημερωθούν με email. ότι μετά τις ψηφοφορίες, ε, στο τέλος των ψηφοφοριών θα συζητήσουμε σύντομα, ε, μετά σύντομο διάλειμμα και μετά θα ψηφίσουμε την... Ε, θα ψηφίσουμε την ένσταση. Θα ψηφίσουμε δηλαδή πρώτα τις, κανονικά τις εκθέσεις για Μακουδάκη, Γκροστέτ κλπ. Και μετά σύντομα στο τέλος θα έχουμε το θέμα αυτό. Ε, καλό διάλειμμα σε όλους για να πέσει το ζάχαρο κιόλας στο αίμα και θα... Ε, ε, ε, θα ξαναπούμε στις 3 η ώρα για την ψηφοφορία.